Good afternoon, ladies and gentlemen. A very warm welcome. I have to send a... Γεια σας, κύριε και κύριοι. Καλώς ορίσατε. Ζητάνε τον συμπαθέ τον κύριο ε, Μπρόκ, αλλά και οι άλλοι αντιπρόεδροι δεν μπορέσαν να βρίσκονται εδώ σήμερα. Οπότε θα πρέπει να υποστείτε εμένα, τον Τσάρλς Τάνοκ. Και για να δούμε τώρα το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Πρώτα-πρώτα έγκριση αυτής. Έχετε κάποια παρατήρηση. Δεν νομίζω. Και μετά έχουμε την έξοδο των πρακτικών τη συνεδρίαση τη 8 Σεπτεμβρίου, τη 6 Οκτωβρίου και τη 10 ε, αλλά και 11 Οκτωβρίου εγκρίνονται γιατί δεν βλέπω ένσταση ούτε παρατηρήσεις. Οπότε τώρα προχωρούμε στο βασικό μας θέμα που είναι η ακρόαση για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή του Σαχέλ. Μεγάλη μου χαρά. Σας εύχομαι καλώς ορίσατε εις αυτή την ακρόαση. Το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ επίκαιρο, ε, σημαντικό και θα το εξετάσουμε από κοινού με την Επιτροπή Ανάπτυξη για να δούμε το τι κάνει, τι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να θίξει και να συζητήσει τι διάφορε προκλήσει αυτή τη περιοχή που έχουν και αρνητικέ επιπτώσει ή στην δική μα ασφάλεια. Και επίση ήμουν εισηγητή για την τελευταία έκθεση του Οκτωβρίου του 2013. Να δούμε επομένω τι αλλαγέ και εξελίξαμε από τότε. Έχουμε συνδυασμό αστάθεια και ανασφάλεια σε ε, αυτά τα σύνορα, ε, ένδια, ε, λοιμό και αυτό πάνω το Σαχέλ. Και οπότε είπαμε ότι υπάρχουν εδώ αδυναμίες και αυτό ήταν έφορα έδαφος για ομάδες ενόπλων, τζιχαντιστές, ε, για την διάδοση εμπορίου όπλων, ε, ε δουλεμπορίας ε, και έχουμε επομένω έτσι έναν διάδρομο από Ανατολή προς Δύση και αντίστροφα της Αφρικής. Στο Μάλι σχεδόν κατέληξε το κράτο το 2012 και έτσι φάνηκε ότι είναι επίγον το να ληφθούν κάποια μέτρα, να βελτιώσουμε και να θωρακίσουμε το Σαχέλ. Και είχαμε τις πρόσφατες τουρκές επιθέσεις στο Μάλι. Οπότε έτσι φάνηκε πόσο ευάλωτη είναι η περιοχή και όπως όλοι ξέρετε ε, προβληματιζόμαστε για την Λιβύη και τη δράση εκεί του Ισλαμικού κράτους. Δεδομένου και των εξελίξεων σε Μοσούλη και Ράγκα. Και επειδή διαφαίνεται ήττα του Ισλαμικού κράτους σε Ιράκ και Συρία, φοβόμαστε μήπως τώρα μεταφερθούν στην Βόρεια Αφρική, μεταφέρουν εκεί δηλαδή τη δραστηριότητά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσπαθεί να διαμορφώσει μια στρατηγική. Αυτό ξεκίνησε το 2011 και αναγνωρίστηκε η περιοχή και είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει μια σφαιρική αντιμετώπιση. Να έχουμε μια στρατηγική για να καλύψουμε την ε, Μαυρετανία, να Φάσο, το Μάλι και τις άλλες χώρες αυτής της περιοχής και έτσι είπαμε ότι μαζί με το Σαγελ έχουμε μια περιφερειακή οργάνωση, φορέα. Θα τα συζητήσουμε σήμερα και έχουμε τον κύριο Άγχελ ε, Λοσάδα, είναι πρεσβευτή, είναι ο πρέσβη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σαχέλ και έχει διαρρομητήσει σημαντικό ρόλο, ούτως ώστε να συντονιστεί ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσέγγιση, για την στρατηγική και επίση και ο κύριο Μέλε, ο οποίο έχει εργαστεί στο Chatham House για το πρόγραμμα τη Αφρική, Ε, κατά σύντοση από τη δική μου εκλογική περιφέρεια για να δούμε τι εξελιξή μου γίνει, τι θέματα υπάρχουν που έχουν σχέση με την ε, σταθερότητα της περιοχής και με μεγάλο ενδιαφέρον επίσης θα ακούσουμε τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι, ε, τι θεωρούν ότι είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί βέβαια χρειάζεται να στηρίξουμε ε, στην περιοχή το, τα κράτη αυτά, τον Νίγερα, το Μάλι. Και, και ο κύριος Βέντα επίσης, ο συνάδελφος είναι ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης. Καλώς ορίσατε. Η Λίντα Μακάβαν δεν μπόρεσε να έρθει, οπότε κύριε Βέντα έχετε τον ε, λόγο. Μπορείτε να μιλήσετε όσο θέλετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας παρουσιάσω μερικά σημεία εξ ονόματος Ανάπτυξης και βεβαίως Προέδρου της κυρίας Λίντα Μάκαβαν. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω και εγώ τους αξιότιμους ομιλητές μας, τον εξούκοτα κύριο Λοσάδα, τον πρέσβη και τον κύριο Πολ Μέρη. Όπως είπατε, η σταθερότητα και η ανάπτυξη της περιφέρειας του Σαχέλ είναι και προς το δικό μας ευρωπαϊκό συμφέρον. Δεν χρειάζεται εδώ να σας θυμίσω ε, τα προβλήματα και τις ανησυχίες που έχουμε με τον φονταμενταλισμό και την τρομοκρατία που αφορά και ε, χώρες ε, ε, του Σαχέλ που είναι το Μάλι, η Νιγηρία και άλλες μακροπρόθεσμα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα γιατί ε, όλα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη σημερινή αστάθεια. οικονομική, ανάπτυξη και κοινωνική σφύριλατη την ειρήνη και την ασφάλεια. Και τη σταθερότητα. Επίση, η σταθερότητα με τη σειρά τη μακροπρόθεσμα οδηγεί σε ανάπτυξη. Οι χώρε Σαχέλ είναι από τι πιο φτωχέ και από τι πιο ευάλωτε του κόσμου. 40 εκατομμύρια είναι οι κάτοικοι ε, που δεν έχουν επιστημιστική ασφάλεια και πάνω από 6 εκατομμύρια χρειάζονται επίγουσα επιστημιστική βοήθεια. Το 2005, 8, 10 και 12 η περιφέρεια εκεί του Σαχέλ γνώρισε τέσσερις επιστημιστικές και διατροφικές κρίσεις. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις και προβλήματα. Πρώτον, ο πληθυσμός εκεί είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος στην κλιματική αλλαγή και στις συνέπειες ε, που... Ε, Έχουμε από τα ακραία καιρικά φαινόμενα με ξηρασίες, πλημμύρες κτλ. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί ε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ζουν από τη γεωργία. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι επηρεάζει και το βιό τους. Στη συνέχεια ο πληθυσμός αυξάνεται με ένα ρυθμό της τάξης του 3%. Μέχρι το 2050 οι 10 χώρες Σαχέλ από την Ερυθρέα ε, ανατολικά μέχρι και τη Σενεγάλη δυτικά θα έχουν πάνω από 330 εκατομμύρια κατοίκους σε σύγκριση με τα 140 που έχουν σήμερα. Όπως γνωρίζουμε, η φυσική πορεία, η γη και το νερό που χρειάζονται για να θρέψουν αυτό τον πληθυσμό σπανίζουν. Αφήστε δε που σήμερα είναι πολύ άνηση η πρόσβαση. 75% του πληθυσμού είναι ηλικία κάτω των 35 ετών και πλήττονται ιδιαίτερα από την ε, ανεργία, από την έλλειψη μόρφωσης, από τη φτώχεια και τον αποκλεισμό. Και πολλοί απογοητεύονται, βλέπουν να ματαιώνονται οι προσδοκίες τους. Και αυτό είναι πρόσφορο έδαφος, αυτό το κενό μπορούν να το καλύψουν ακραίες ομάδες. Ορισμένοι αποφασίζουν να μεταναστεύσουν από τους νέους αυτούς για να βρουν την τύχη τους αλλού. Ε, Στι περισσότερε περιπτώσει είναι σε άλλε Ευρω... Ε, αφρικανικέ χώρε και ορισμένοι έρχονται και στην Ευρώπη. Βεβαίω, ο πόλεμο και η πολιτική ασφάλεια στο ε, Μάλι, στη Λιβύη και την Νιγηρία εντείνουν το πρόβλημα και έτσι εκτοπίζει το πληθυσμό από τη μία χώρα στην άλλη. Είμαι βέβαιο ότι θα ακούσουμε και θα μάθουμε περισσότερα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, αλλά θυμίσω μερικά στοιχεία. Είμαστε από τους μεγαλύτερους δωρητές και ανθρωπιστικής βοήθειας και γενικότερα. Πάνω από 200 εκατομμύρια έχουμε δώσει ε, σε 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν πρόβλημα ε, υποσυτισμού. Και αυτό είναι το 1 τέταρτο όλων των αναγκών των διατροφικών και πάνω από 43% ε, του παιδικού υποσυτισμού. Υπάρχει μια πρωτοβουλία για το Σαχέλ των Ηνωμένων Εθνών, μια διεθνή συμμαχία για να μειωθεί ε, ο χρόνιος υποσυτισμός και να φτάσουμε ε, το 2032 ε, στην εξάλληψη του υποσυτισμού. Όλα αυτά, είπαμε, είναι αρνητικοί παράγοντες και οδηγούν τον κόσμο στη μετανάστευση. Ε, έχουμε και προγράμματα που έχουμε συμφωνήσει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη, επίση μακροπρόθεσμα. Ε, ταυτόχρονα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα προγράμματα είναι καλά, αλλά δεν είναι πλήρη ε, ούτε επαρκή. Στρατηγικέ υπάρχουν διάφορε για τη Σαχέλ, μάλιστα περισσεύουν κιόλα. Αυτό που λείπει είναι οι διαφορετικέ αυτέ στρατηγικέ να συγκεντρωθούν και να ε, καταλήξουμε σε κάτι πιο συνεκτικό και αποτελεσματικό για όλη την περιοχή. Με διεθνή ε, συμμετοχή, τοπική, περιφερειακή και βεβαίω των ίδιων των ενδιαφερομένων. Η δική μα στρατηγική και η δράση μα για το Σαχέλ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και Αφρικανούς πέραν του Σαχέλ, δηλαδή την ΕΚΟΒΑΣ για παράδειγμα και την Αφρικανική Ένωση και να έχουμε υπόψη μας και την κατάσταση στη Βόρεια Αφρική. Αξίζει λοιπόν να αναφέρουμε ότι του χρόνου το 2017 ε, αναμένεται ε, να ε, εγκριθεί μια νέα Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη, μια νέα στρατηγική για την Αφρική και να δούμε πώς θα πλαισιωθεί συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ μετά τη λήξη ε, του Κοτονού το 2020. Πριν τελειώσω, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, προβλέπει το Φεβρουάριο 2017 δύο ε, αποστολές, μία στη Σενεγάλη, για να καταλάβουμε καλύτερα τη δυναμική της μετανάστευσης και πώς υπάρχει συνεργασία για τη διαχείριση αυτής, και μια δεύτερη αποστολή πάλι το Φεβρουάριο στο Τσάτ, έτσι ώστε να αναλύσουμε τις ε, περίπλοκους δεσμούς ανάμεσα στην ε, αστάθεια των κρατικών ε, δομών, τη φτώχεια, την βεβαιότητα, τον πολιτικό εξτρεμισμό. Ελπίζω η σημερινή ακρόαση να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και αναμένω. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα εισαγωγικά σχόλια από αναπτυξιακή σκόπια και θα δώσω τώρα ε, ε, το λόγο ε, στον κύριο Άγγελο Μέντες για να κάνει τη δική του παρουσίαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Βέντα. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη μου τιμή που ήρθα αλλά και μεγάλη ικανοποίηση, γιατί για δεύτερη φορά εδώ πέρα είμαι στην υποεπιτροπή σας, γιατί είχα πάει και στην υποεπιτροπή της Άμυνας και αν δεν έχετε πρόβλημα, άλλο να σα τα πω και στην Λίγκο Φράγκα τη περιοχή, δηλαδή τα γαλλικά. Σα ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου τιμή το ότι με καλέσετε σήμερα εδώ. Μιλούμε για μια εξωτερική πολιτική προ το Σαχέλ. Και το Σαχέλ, όπω πάρα πολύ σωστά αναφέρθηκε προηγουμένω, έχουμε 12 χώρε. Αυτό, έτσι ορίζεται το Σαχέλ και ε, όλε αυτέ βρίσκονται σε απόσταση τριών ωρών με το αεροπλάνο Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε η ασφάλεια αυτών των χωρών είναι 100% και η δική μα ασφάλεια. Και αυτό είναι η αφετηρία, αυτό είναι η βάση από την οποία αρχίζει η προβληματική μα. Είναι τελικά τα σύνορα στα σύνορά μα. Είναι αυτοί που λένε ότι είναι προκεχωρημένε θέσει των σύνορων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε με δεδομένη την κρίση σήμερα στη Λιβύη, όλοι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι με δεδομένο το κενό που υπάρχει στη Λιβύη ουσιαστικά ε, εκεί είναι το σύνορό μας. Και ακριβώς όπως προσπάθησα να, <clears throat> να σας πω. Οπότε χρειάζεται να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Και ε, λέμε ότι η ασφάλεια τους είναι δική μας ασφάλεια όταν μιλούμε για Σαγέλ. Πώς όριζε το Σαγέλ για να δούμε ε, σε, σε τρεις άξονες πώς έχει κατάσταση. Πρώτα-πρώτα, ο ορισμός είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα ακαδημαϊκό, πανεπιστημιακό. Σύμφωνα με τον ορισμό που έχουμε, Έχουμε την κατανομή σε διάφορε χώρε αυτή τη περιοχή, ή τόσο τι χώρε περιλαμβάνει, και δεύτερον να δούμε ποια είναι η στρατηγική και το, το, το πρόγραμμα περιφερειακή δράση. Και κατά τρίτον, ο τρίτο άξονα που θα συζητήσουμε είναι το μέλλον της στρατηγικής. Και θα έχουμε ως βάση δύο στοιχεία. Πρώτα-πρώτα τη διαδικασία ειρήνευση στο Μαλί και την περιφερειοποίηση με το G5 και την ε, πολιτική που τώρα έχει χαράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί επομένως είναι οι τρεις βασικοί άξονες που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Πρώτα-πρώτα η έννοια. Αναμφίβολα η κρίση του Σαχέλ είναι μια κρίση περιφερειακή. Αυτό δεν χωρεί καμιά συζήτηση και άρα θα πρέπει να δώσουμε τον ορισμό αυτής της περιοχής, της περιφέρειας, ε, γιατί πάνω σε αυτό θα εφαρμόσουμε τα όσα θα αποφασίσουμε. Έχουμε τρεις διαφορετικές έννοιες που καλύπτει η λέξη, ο όρος Σαχέλ. Πρώτα-πρώτα γεωγραφικά, δεύτερον θεσμικά και τρίτον γεωστρατηγικά. Πρώτα-πρώτα από πλευράς γεωγραφικής. Είναι απλό. 5.700 χιλιόμετρα. Σαχέλ ε, σημαίνει όχθη, άκρη. Άρα πρόκειται για τη ζώνη από Ερυθρά θάλασσα μέχρι τον Ατλαντικό και διασχισμένο αυτό ο όρο, αφορά αυτό ο χώρο 12 χώρε που έχουν γίνει χαρακτηριστικά. Το ίδιο επομένω ισχύει και για την θεώρηση των πραγμάτων πλευρά ασφάλεια, ανθρωπιστική, διακυβέρνηση, ακόμα και όσον αφορά το κλίμα. Σημαντικό και αυτό. Αλλά επίση βεβαίω υπάρχουν και εκείνα χαρακτηριστικά για ασφάλεια και μετανάστευση. Αυτά από πλευρά γεωγραφική. Δεύτερη πτυχή του θέματο είναι η θεσμική πτυχή. Γιατί μιλούμε για θεσμική άποψη θέματος, γιατί μιλούμε για πέντε χώρες. που βρίσκονται γύρω-γύρω από τον ε, Νίγηρα και εκεί έχουν ξεκινήσει ε, κάποιοι πάρα πολύ αρχαίοι ε, πολιτισμοί όπως το, του Τιμπουκτού, του Γκάου και γύρω από αυτό τον ποταμό βρίσκονται αυτές οι χώρες και μαζί με Τσάδ και Μαυριτανία θέλαν να συμπίξουν την πλατφόρμα G5 που ξεκινούν από μια απόφαση, απόφαση αρχηγών κρατών. Κυρίαρχη απόφαση ούτως ώστε να έχουν αυτή την πλατφόρμα για κοινέ σχέσεις, για πολιτική ανάπτυξη και ασφάλειας. Αυτό θέλαν να συμπίξουν αυτές οι χώρες. Πρόκειται για μια ένωση κρατών επομένω. 19 12 του 14 έγινε αυτό. Και τώρα υπάρχει μια μόνιμη γραμματεία. Στο Νουαρσότ, στην Μαυριτανία είναι η έδρα, υπάρχει κυκλική εναλλαγή και επίσης εμπλέκεται και το Τσάδ. Οπότε θα ασχοληθούμε και με αυτή την πλατφόρμα, αυτό το θεσμικό όργανο. Τρίτο στοιχείο τώρα, το οποίο είναι η γεωστρατηγική υφή. Ξεκινούμε από αυτό το G5 το οποίο συγκροτήθηκε για να αναλύσουμε μια κρίση η οποία βεβαίω έχει αντίκτυπο και στην κρίση της Λιβύης. μία κρίση τέλο πάντων ε, συμπαρασύρει και την άλλη και στην ε, Νιγηρία με την Μπόκο Χαράμ και επομένως όλα αυτά παροξύνουν την κατάσταση. Αυτό λοιπόν πλευρά τη Επίση, Επίσης, δεύτερο επίπεδο σε αυτή τη γεωστρατηγική θεώρηση είναι οι χώρε του Σαχέλ, Είναι αυτέ οι χώρες, οι του Σαχέλ. Ε, δεν μπορούμε να, πούμε, δηλαδή, να βγάλουμε έξω από το Σαχέλ την, ε, τη Βόρεια Νιγηρία ή την Σενεγάλη για παράδειγμα. Όμως θεωρούμε ότι η καρδιά της περιοχής είναι το G5. Όμως και η Αλγερία και η Σενεγάλη και η Νιγηρία ε, και αυτοί επομένω έχουν ε, πλησιάσει το G5. Οπότε αυτές οι χώρες λόγω των αδυναμιών, των θεσμικών και πολιτικών που έχουν κάπως τις εξομοιώνουμε με τις χώρες αυτές το G5, τις κυρίως χώρες του Σαχέλ. Είναι σημαντικό πάντως τώρα να δούμε τη δεύτερη θεώρηση των πραγμάτων, τη θεσμική και τη γεωστρατηγική. Άρα θα πρέπει να έχουμε πιο άμεση ε, παρέμβαση σε αυτό το επίπεδο και επίσης να λάβουμε υπόψη και την τρίτη πλήτη γεωστρατηγική όσον αφορά τις αποφάσεις που οφείλουμε να πάρουμε. Γιατί όπως είπαμε δεν μπορεί να γίνει τίποτα στο Σαχέλ, να λάβουμε υπόψη η Ιγυρία και η Αλγερία, αλλά να λάβουμε επίσης υπόψη την ΣΕΝΤΕΟ αλλά και την Αφρικανική Ένωση. Όμως επίσης Έχουμε και άλλες δύο σημαντικές ε, περιοχές οι οποίες επηρεάζουν το Σαχέλ. Πρόκειται για το Μαγρέμπ αλλά επίσης και την Δυτική Αφρική. Επομένως και εδώ υπάρχει θέμα, έχουν σημασία αυτές οι περιοχές για τη μετανάστευση και φυσικά ε, οι συνέπειες βρίσκονται επί των χωρών προορισμού που είναι δηλαδή η Ευρώπη. Θα πρέπει επομένω να λάβουμε υπόψη όλε αυτέ τι έννοιε για να μπορέσουμε να έχουμε μια συγκεκριμένη και άμεση πολιτική για το Σαχέλ. Πάει αυτό. Δεύτερον, η στρατηγική. Η στρατηγική τη Ευρώπη για το Σαχέλ και επίση το πρόγραμμα δράση σε περιφερειακό επίπεδο. Η στρατηγική. Α ε, δεχθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ε, πρώτη στο να έχει τη σχετική στρατηγική. Γιατί υπάρχουν πολλές στρατηγικές που αφορούν το Σαχέλ. Δεν είναι κακό αυτό γιατί όσο πιο πολλές στατικές έχουμε περισσότερο καταδεικνύεται το ενδιαφέρον της, της διεθνούς κοινότητας. Άρα θα πρέπει να υπάρχει όμως σωστή, σωστό, σωστή, συντονισμός μεταξύ αυτών των ε, πολιτικών. Άρα έτσι προκύπτει κάτι θετικό από τις διαφορές, δικές, πολλές στατικές. Επομένως, η στρατηγική θα πρέπει να έχει δύο πυλώνες την ασφάλεια και όπως είπε ο κύριος Βέντα την ανάπτυξη. Δεν μπορεί να υπάρχει ασφάλεια χωρίς ανάπτυξη ούτε ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια και όλα αυτά θα πρέπει να υπήκουν στις ε, αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία την ε, προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Αλλά ασφάλεια και ανάπτυξη είναι οι βασικοί πυλώνες. Αλλά και το στοιχείο της ε, ασφάλειας ε, βεβαίω είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Γιατί είπαμε, ο ένας πυλώνας εξαρτάται από την ύπαρξη του άλλου. Με βάση αυτή τη στρατηγική τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρεξε τέσσερις κατευθυντήριες γραμμές δράση. Όπως είπαμε, αυτά ξεκίνησαν το 2011. Πρώτη δράση αφορά την ανάπτυξη χρηστή διακυβέρνηση, αλλά επίσης και την επίλυση των ε, διαφορών και συγκρούσεων. Και αυτά γίνανε, ισχύουν και για την κρίση του Μαλή. Εκεί κατέβαλε προσπάθειε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, τις ε, ειρηνευτικές, υπεγράφησαν από τον προκατοχό μου. Ήμασταν εμεί επομένω οι εγγυητέ, αλλά και στη συνέχεια και παρακολούθηση των εξελίξεων μέσω τη υπηρεσία μα έχουμε συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία εποπτείας και παρακολούθηση. Άρα, ανάπτυξη, χρηστή διακυβέρνηση και επίλυση των ε, συγκρούσεων. Και για την ανάπτυξη, όπως αναφέρθηκε, εμείς είμαστε ο βασικός ε, δανειστής, ο βασικός ε, σπόνσορας μιλούμε για 3,5 εκατομμύρια ευρώ για το Σαχέλ, αλλά επίσης υπάρχουν και εθνικά προγράμματα. Η δεύτερη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αφορά την διπλωματία αλλά και την πολιτική. Οπότε σε αυτό το επίπεδο έχουμε την ε, πολιτική υποστήριξη σε αυτό το G5. Πάνω από 17 αποστολές έχω κάνει τελευταία χρονιά, ούτως ώστε να δούμε τι γίνεται με μια κοινή στατική αυτών των πέντε χωρών για να υλοποιηθεί αυτό το στρατηγικό όραμα που έχουν ανακοινώσει οι ηγέτες τους. Τι μπορούν να κάνουν αυτές οι ίδιες οι χώρε, διπλωματικά και πολιτικά. Εκεί προβάλλεται και δράση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βασικός εισφορέας και δωρητή είναι το πιο σημαντικό. Οπότε και μπαίνουμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία της περιφερειοποίησης που είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστεί και ως τρίτο στοιχείο, ως τρίτη δράση είναι ασφάλεια και κράτος δικαίου. Όπως είπαμε είναι βασικός ο πυλώνας της ασφάλειας. Ήταν καθηγητήρια γραμμή που εγκρίθηκε όταν ε, χαράθηκε αυτή η στρατηγική και έχουμε εκεί κάποια αποστολή, η ΚΑΠ για το Μαλί και τον Νίγηρα. Συμβάλλουμε στην ε, οργάνωση αστυνομία, στην ΕΤΕΜ επίσης για εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων στο Μαλί. Θα τα συζητήσουμε περαιτέρω, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε το ότι υπάρχει σημαντικό έργο που γίνεται από αυτές μας τις ε, αποστολές. Επίσης προσπαθούμε να αναδιαρθρώσουμε ε, τις διοικητικές αρχές ε, της ε, δύναμης ασφαλείας αυτών των χωρών. Επομένως δίνουμε προτεραιότητα όσον αφορά τον εξτρεμισμό, όσον αφορά τη ριζοσπαστικοποίηση και όλα αυτά θα τα το πρόγραμμα δράσης. Και για αυτές τις στρατηγικές πώς θα δούμε τι θα γίνει με την κρίση στο Μαλί. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να συμμετάσχει 100% σε όλες τις ε, κινήσεις υλοποίησης της διαδικασίας του Αλγερίου για το Μαλί. Αλλά ε, Επίση με την αποστολή μας προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες, δεν αρκούν όμως αυτά. Οπότε το 2015, συγκεκριμένα τον Απρίλιο, εγκρίθηκε και αποφασίστηκε αυτό το πρόγραμμα δράσης περιφερειακού επίπεδου, το οποίο έχει τέσσερις άξονες και οι προτεραιότητες. Υιοθετεί ουσιαστικά αυτές τις γραμμές, αλλά είναι πολύ πιο συγκεκριμένες οι προτεραιότητες που έρχονται να απαντήσουν σε μια πολύ συγκεκριμένη συγκυρία κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής κρίσης και μετά της κρίσης με τα θέματα ασφαλείας που είδαμε στο Σαχέλ στην καρδιά του και στη Σαχάρα. Θυμάμαι κάτι που είχε αναφέρει ο Υπουργό Μπαζούν που είναι τώρα Υπουργό Εσωτερικών στον Ήγηρα και έλεγε ότι για εκείνου η Σαχάρα ήταν σε μια προστατευτική ασπίδα και αισθάνονταν άνετα μέχρι που ξέσπασε κρίση στη Λιβύη. Έκτοτε η Σαχάρα είναι για μα, λέει η πηγή όλων των συγκρούσεών μα γιατί δεν την ελέγχουμε. Άρα θα χρειαστούν βοήθεια και πλαισίωση και το κάνουμε ήδη σε τέσσερι προτεραιότητε, όπω σα είπα. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η καταπολέμηση τη ζήσεως Τι κάνουμε προ την κατεύθυνση αυτή. Κατά κύριο λόγο, έχουμε καταρτήσει ένα ε, ερωτηματολόγιο και το έχουμε στείλει σε όλες τις αντιπροσωπείες και στις πέντε χώρες, τις δικές μας, για να δούμε πώς έχει ζωστικοποιήσει και πώς ε, την ε, καταπολεμόμουν. Και το G5 το υποστηρίζουμε, κάνουν διάφορα σεμινάρια εκεί και καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα, σε κάποια ενδεικτικά σημεία κυριαρχεί ένα πολύ λεπτό και ευαίσθητο θέμα και για σας πιστεύω. Είναι το θέμα του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους. Αυτό που στα γαλλικά λέγεται λαΐσιτε. Μπορεί να είναι ταμπού αυτό, αλλά στην Αφρική έχει και μια άλλη διάσταση. Ε, σημαίνει ότι δεν αναμειγνύεται το κράτος ε, στα, της θρησκείας αλλά αυτό ε, αφήνει ένα κενό το οποίο έρχονται να πληρώσουν αμέσω οι τζιχαντιστέ. Θα πρέπει να το συζητήσουν γιατί αυτό έχει να κάνει με τον έλεγχο ή το μη έλεγχο των ημάμιδων ή των χρηματικών ροών που χρηματοδοτούν τα ντεμένη και τα τζαμιά ή το θέμα τη εκπαίδευση, κατάρτιση θρησκευτική των ημάμιδων ή να υπάρχει ένα πλήρη κατάλογο όλων των τζαμιών, όλων των ημάμιδων και να ξέρουν τι υπάρχει. Ε, αυτό τώρα ε, ξεκινάει ως προσπάθεια των χωρών αυτών των πέντε και θα πρέπει και εμείς να τους βοηθήσουμε και προσπαθούμε να το κάνουμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν, καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης είναι το πρώτο στοιχείο του περιφερειακού προγράμματος δράσης. Το δεύτερο που συνδέεται άρρηκτα με το προηγούμενο είναι το εξή. Οι νέοι, τι γίνεται με την νεολαία. Αυτό είναι ένα θέμα που επανέρχεται και το είπε και ο κύριος Βέντα, έχει να κάνει με ε, τη δημογραφική έκρηξη ε, που συντελείται ε, ήδη και σήμερα. Πραγματική έκρηξη είναι αυτή και αν θέλετε και ορολογιακή βόμβα και βραχυπρόθεσμα. Θυμάμαι τον πρόεδρο Ισούφου, τον πρόεδρο του Νίγηρα, μου έλεγε πάρα πολύ πρόσφατα ότι η χώρα του έβλεπε το πληθυσμό της να διπλασιάζεται στο παρελθόν κάθε 30 χρόνια και σήμερα κάθε 18 χρόνια. Κάθε 18 χρόνια έχουμε άλλον έναν νίγηρα πληθυσμιακά. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει. Προσπάθησαν να προχωρήσουν σε έλεγχο, όχι ακριβώς σε έλεγχο γεννήσεων, αλλά κάποια προγραμματισμό οικογενειακό, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχουν θέματα θρησκευτικά εκεί και πολιτισμικά. Αλλά γνωρίζουν ότι είναι μέγα πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίζουν. Και είπατε εκπρόσωπο από δική μα πλευρά, η κυρία Μογκερίνη, την τελευταία φορά που συνεδρίασε με ε, του υπουργού του G5 των εξωτερικών, αναφέρθηκε στο περιθώριο αυτή τη συνεδρίαση. έκανε μια άλλη εκδήλωση με του νέου του Σαχέλ και συνεχίζεται αυτό. Εγώ προσπαθώ να επισκέπτομαι τις χώρες αυτές για να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο μεταξύ της νεολαία των κρατών αυτών για να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα, η συνεργασία, να υπάρξει μια πραγματική ένωση των πέντε κρατών. Αυτό το στοιχείο της ε, νεολαίας είναι από τα πιο σημαντικά. Υπάρχει μια πλατφόρμα του G5 για τους νέους, την οποία παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή. Ο δρόμος των νέων στο Σαχέλ ονομάζεται αυτή η πλατφόρμα και την ε, συνέστηση τι εκπρόσωπος. Αυτή ήταν η δεύτερη προτεραιότητα. Τρίτη προτεραιότητα, θα την ξέρετε κι εσείς αλλήμωνο, μετά τα όσα συνέβησαν, είναι το θέμα της μετανάστευσης. Μετανάστευση και κινητικότητα. Συμπεριλαμβάνεται αυτό ρητά στο περιφερειακό πρόγραμμα δράσης. Η μετανάστευση, γνωρίζουμε όλοι, μετά τη συνεδρία στη Βαλέτα της Μάλτας και μετά τις τρομερές σκηνές που βλέπουμε στην τηλεόραση, οδήγησε σε τεράστια αλλαγή τι έχουμε τώρα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη η στιγμή και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, χωρίς καμιά αμφιβολία. Ένα καταπίστευμα, 1,8 δις και 1,1 ειδικά για το Σαχέλ. Υπάρχουν διάφορα έργα λοιπόν που έρχονται να αντιμετωπίσουν τις βαθιές αιτίες τη ρίζα τη Αυτό έχει να κάνει με την ανάπτυξη, με την νεολαία, ε, με την ε, αντίσταση ε, και την αφεκτικότητα μιας κοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα λαμβάνει αυτά υπόψη και έχουμε ως παράδειγμα την πόλη Αγκαντές στο Νίγηρα και προσπαθήσαμε να φτάσουμε ε, ω εκεί σε αποκεντρωμένη προσπάθεια γιατί είναι συμβολική για τη μετανάστευση η πόλη αυτή Αγκαντές από τον Ήγηρα. Αυτή ήταν η τρίτη προτεραιότητα και έρχομαι στην τέταρτη που συνδέεται και με τις προηγούμενες. Αυτό είναι ο έλεγχος και η διαχείριση των συνόρων. Θέλω να επιμείνω σε αυτό το στοιχείο. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι υπάρχει μια προστιθέμενη αξία του G5. Τι σημαίνει αυτό. Αυτές οι πέντε χώρες ε, ενώνονται και δρούν για ένα θέμα που είναι από τα πιο δύσκολα, η διαχείριση των συνόρων. Γιατί αν δεν μπορούν οι χώρε αυτέ να ελέγχουν τα σύνορά του, θα συνεχίζεται η διακίνηση, παράνομη, η λάθρομετανάστευση, ε, εγκληματικά δίκτυα που θα αλωνίζουν εκεί. Με διάφορα προβλήματα, εγκάρσια, οριζόντια και κάθετα και η απάντηση είναι μόνο περιφερειακή. Δεν μπορεί να είναι διαφορετική. η Ευρωπαϊκή Ένωση το θέτει αυτό με τρόπο πάρα πολύ συγκεκριμένο και ρητό. Τώρα θα μου πείτε, ωραία όλα αυτά, τι εργαλεία έχουμε για να εφαρμόσουμε αυτές τις πολιτικές. Ε, τα έθιξα προηγουμένω. Δύο ειδών είναι κυρίως. Χρηματοδοτικά μέσα και θεσμικά εργαλεία. Τα χρηματοδοτικά ποια είναι. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι πάνω από 12-13% που πηγαίνουν στο Σαχέλ και με άμεση μακροοικονομική βοήθεια για κάποιες από αυτές τις χώρες. Ξέρετε, όλοι οι πρόεδροι των κρατών ζητούν ε, την άμεση ενίσχυση και όχι μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης. Είναι πιο εύκολο για αυτούς και πιο δύσκολο να ελεγχθεί. Αλλά ε, με την κρίση που γνωρίζουμε, στον Ήγηρα έχουν ένα πρόγραμμα ανάπτυξης που είναι τα τρία εν στα γαλλικά. Οι Νιγηριανή... Ε, ε, τρέφουν τους Νιγηριανούς, les ε, έχουν αφιερώσει ε, πάρα πολλά κονδύλια, το 1 τρίτο περίπου, για την ασφάλεια και για την αντιμετώπιση του Μποκο Χαράμ. Έχουμε λοιπόν χρηματοδοτικά μέσα, αλλά και θεσμικά, όπως σας είπα προηγουμένως. Και ποια είναι τα θεσμικά, αναφέρθηκα. Είναι οι δικές μας αποστολές εκεί UCAP ε, Νίγηρας, UCAP Μαλή, ε, ATM Μαλή ή UTM Μαλή. Αυτή είναι η άμεση δράση, θα λέγαμε, επιτόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τόσο της ασφάλειας όσο και τα υπόλοιπα για να έρθει η ε, ανάπτυξη που ελπίζουμε. Άλλο θεσμικό εργαλείο είναι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης και το γραφείο μου το ίδιο. Όπως σας είπα, πάνω από 20 φορές μέσα σε 10 μήνες ε, χτενίσαμε την περιοχή εκεί και προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε και τα ευρωπαϊκά κράτη για τη σημασία όλων αυτών. Που σας είπα ότι η ασφάλεια του Σαχέλ σημαίνει ασφάλεια και για την Ευρώπη. Είδαμε λοιπόν ποια ήταν η στρατηγική μας, ποιο είναι το πρόγραμμα δράσης. Ένα τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να τονίσω, κύριε Πρόεδρε. Και δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη σε σχέση με τη δική σας έκθεση, αν είναι θετική ή αρνητική εξέλιξη λοιπόν. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο ζητήματα εδώ. Την ευτική διαδικασία στο Μάλι πρώτα και μετά την περιφερειοποίηση γενικότερα ευτική διαδικασία. Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι έχουμε προχωρήσει. Βέβαια, είχαμε καθυστερήσεις, αλλά καμιά φορά βιαστήκαμε και υπερβολικά. Είναι περίπλοκη η κατάσταση και η κυβέρνηση βασίζεται σε μια στρατηγική που λέει δεν ε, κάνω τα βήματα προς την κατεύθυνση την πολιτική εφόσον δεν έχω εξασφαλίσεις από τους του ΕΡΕΚ. Και το αντίθετο λένε οι του ΕΡΕΚ. Δεν έχουμε την πολιτική στήριξη, αλλά δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε την ασφάλεια της περιοχής. Παρά τις πολλές επικρίσεις κατά της ενευτικής διαδικασίας, η οποία αποτελματώνεται, δεν το αρνούμε, έχουμε δύο πολύ σημαντικές πρόοδους. Πρώτον, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει ρόλο εκεί. Ουδής δεν μιλά για παραβίαση της εδαφικής αγκαιρεότητας στο Μάλι. Ενώ πριν από τρία χρόνια ε, δεν το έλεγαν μόνο ως ενδεχόμενο, ε, θεωρούσαν ότι το Βόρειο Μάλι θα μπορούσε να αποσχιστεί. Ε, κανείς σήμερα δεν αφισβητεί την εδαφική αγκαιρεότητα, επαναλαμβάνω. Και μετά όλα αυτά τα κινήματα που μέχρι πριν από λίγους μήνες, μέχρι πριν από δύο χρόνια, άλλοι σκοτώνονταν και ε, ε, πολεμούσαν, βρίσκονται γύρω από το ίδιο τραπέζι σήμερα ε, σε μια ενευτική διαδικασία και διαπραγματεύονται με μια επιτροπή παρακολούθησης των συμφωνιών που συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η επιτροπή και αυτή η διαμεσολάβηση στην οποία συμμετέχουμε είναι κάπως προβληματική γιατί είναι πολύ ενεχόμενη αλλά προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να προχωρήσουμε. Αν έχετε ερωτήσεις για την ευτική διαδικασία, με χαρά να απαντήσω. Δεν θέλω να, παραμείνω, να επιμείνω σε πολλές λεπτομέρειες τώρα. Η δράση μας λοιπόν είναι και στα πλαίσια ε, του ΟΗΕ, γιατί το ψήφισμα 2295 του Συμβουλίου Ασφαλείας μας δίνει εντολή ε, σε μένα και στην ε, ομάδα μου και στο επιτελείο να συνεργαστούμε με το Μαλί για την αναδιάρθρωση των δυνάμεων ασφαλείας. Αυτά για την ευτική διαδικασία. Ένα δεύτερο στοιχείο όπου υπάρξει, έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος είναι η περιφερειοποίηση. Τι θα πει αυτό. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα νέο στάδιο. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πέντε χώρες του Σαχέλ, το G5. Έχουμε περάσει μια επιχειρησιακή φάση. Δεν βρισκόμαστε στο σχεδιασμό ή στο στήσιμο της συνεργασίας. Υπάρχει αυτή. Η συνεργασία είναι γεγονός επιτόπου. Έχουμε ενισχυμένο διαρθρωμένο διάλογο με ε, οδικό χάρτη και φύλλο πορείας και όπως είπε ο κύριος Βέντα, ανάγκη συντονισμού. Το πρώτο στοιχείο είναι αυτός ο ενισχυμένος και διαρθρωτικός διάλογος ε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πέντε κρατών. Η κυρία Μογκερίνη συμμετέχει εκεί στη Συνόδος κορυφής και μάλιστα την τελευταία φορά ε, έλαβε χώρα τον Νοέμβριο αυτή πέρυσι στη Τζαμένα του Τσάντ. Επιπλέον, σε υπουργικό επίπεδο γίνονται συνεδριάσεις συμμετέχει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και όλοι οι Υπουργοί Εξωτερικών του G5 παρουσία της κυρίας Μαγκερίνη και εγώ προσωπικά συμμετέχω ε, σε όλους τους σχηματισμούς, ε, ασφάλεια, ε, μετανάστευση, νεολαία κτλ. Αντίστοιχα, υπάρχει ένας μόνιμος γραμματέας του G5 που συμμετέχει στις δικές μας συνεδριάσεις. Την περασμένη εβδομάδα τον συνέστησα στο ΚΟΠΣ, στην επιτροπή αυτή που μίλησε και μάλιστα σε μια συνεδρίαση για την ασφάλεια στο Βερολίνο. Δηλαδή, είναι καλά διαρθρωμένος, εγκατεστημένος ο διάλογος, εδρεωμένος, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται δικός χάρτης, τον οποίο και εγκρίναμε ε, και έρχεται να κάνει τον απολογισμό κάθε φορά που βρισκόμαστε και τι θέλουμε να κάνουμε, πού θέλουμε να πάμε. Είναι γεγονό ότι ο τομέας της ασφάλειας στο G5 είναι εκείνος ο οποίος έχει προχωρήσει περισσότερο. Δεν ε, χωρά καμία αμφιβολία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στη χρηματοδότηση άμεσα ε, ε, χρηματοδότηση εμπειρογνωμόνων για την ασφάλεια και την άμυνα ε, και στην Τζαμένα στην Προεδρία του G5. Επίσης συμμετέχουμε σε όλες τις εργασίες τους και χάρη στο καταπιστευματικό ταμείο πρόσφατα εγκρίναμε τρία έργα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ασφάλεια. Επαναλαμβάνω και ζητώ συγγνώμη που σας κουράζω ε, που επαναλαμβάνομαι, αλλά όταν υπάρχει κενό εξουσίας, όταν υπάρχει κενό κρατικής ε, υπόστασης, αυτό είναι το οξυγόνο για την τρομοκρατία. Όπου υπάρχει κενό εξουσίας θα πρέπει να καλυφθεί, αλλιώς θα το καλύψουν κάποιοι άλλοι. Θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτεται. Γι' αυτό υπάρχει το πρόγραμμα ε, ΠΑΣΕΚ που ε, χρηματοδοτείται από το καταπίστευμα, ε, ενισχύει ε, το κέντρο ε, του Μάλι. Υπάρχει ένα project που λέγεται Γκάρσι και συμμετέχει η γαλλική χωροφυλακή, η ισπανική, η ιταλική για την εκπαίδευση των αστυνομικών δυνάμεων. Και ένα τρίτο στοιχείο αυτού του οδικού χάρτη που προχωρεί καλά και το προωθούμε είναι το θέμα του συντονισμού που ανέφερε και ο κύριος Βέντα. 16 στρατηγικές έχουμε, μάλιστα 17 τώρα έχουν γίνει για το Σαχέλ, πολλές είναι βέβαια. Καλά είναι, αλλά είναι πολλές. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Στις 29 Νοεμβρίου θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί στην Τζαμένα σε μια στρατηγική πλατφόρμα και θα συμμετέχουν όλοι. Ε, η Οικονομική Κοινότητα Δυτικοαφρικανικών Κρατών, η Αφρικανική Ένωση, ο ΙΕ κτλ. Έτσι ώστε να υπάρχει μια πολύ στενή σύνδεση με την Αφρικανική Ένωση πρώτα απ' όλα, γιατί καμιά φορά εκεί υπάρχει πρόβλημα. Πώς να το πω τώρα. Η Αφρικανική Ένωση δεν αντιλαμβάνεται πάντα πολύ καλά τι συμβαίνει στις πέντε χώρες του Σαχέλ. Αυτό τώρα έχει, έχει ε, αλλάξει. Ε, υπάρχει στο Νουαξότ ε, μια τοπική παρουσία του ΟΗΕ που αναγνωρίζει το G5 ως οντότητα, γιατί η Αφρικανική Ένωση δυσκολεύεται ακόμα να το αναγνωρίσει. Υπάρχει η Μίνουσμα, η αποστολή του ΟΗΕ στο Μαλί, δεν μίλησα πολύ γι' αυτό, θέλετε με χαρά να επεκταθώ. Ε, υπάρχει η αποστολή Μπαρκάν η γαλλική που έχει τεράστια απήχηση και ε, πραγματικά επέτρεψε να συγκρατηθεί η τεράστια έκρηξη που θα μπορούσε να έχει σημειώσει ο τζιχαντισμός εκεί στην περιοχή. Αυτά ήταν οι τρεις μεγάλοι άξονες, δεν ξέρω μήπως μακρηγόρησα πάρα πολύ, αλλά γιατί τα λέω αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής, δεν χωρά καμία αμφιβολία, αλλά χρειαζόμαστε να είμαστε και ορατοί, να ε, είμαστε προβεβλημένοι. Το κάνουμε σε συνεργασία με τους G5, τις πέντε χώρες περιοχής, αλλά πάντα αυτό που μας διέπει είναι να γίνει κτήμα τους, να έχουν εκείνη την ιδιοκτησία, όπως λέμε, αυτών των πραγμάτων. Οι ίδιες οι χώρες Σαχέλ δεν θα έρθουμε εμείς να τους επιβάλλουμε. Εμείς τους βοηθάμε, τους πλαισιώνουμε, τους συνοδεύουμε. Και ε, καταλήγω με κάτι που έχει μπει Φεντερίκα Μογκερίνη και το επαναλαμβάνουμε συχνά, αλλά είναι πολύ καλό ως σύνοψη. Εμείς δεν εργαζόμαστε για την Αφρική, εργαζόμαστε μαζί με την Αφρική, συνεργαζόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρέσβη για αυτήν την ε, πολύ περιεκτική παρουσίαση όλων των ε, πτυχών ε, της ασφάλειας, της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας, των συνοριακών ελέγχων αλλά και των διαφορών αποστολών από την πλευρά μας, τη σχέση λοιπόν όλων αυτών και βέβαια αυτό μας δείχνει ακριβώς το πόσο περίπλοκη είναι η συνοπτική ε, εικόνα και βέβαια μας ε, κάνατε και μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση σε ό,τι αφορά το G5 που υπάρχει εδώ και τρία χρόνια ε, και βέβαια γνωρίζω πως κάποια από τα σύνορα εδώ των χωρών πραγματικά βρίσκονται στα σύνορα της ίδιας της ερήμου οπότε εκεί πραγματικά η όλη προσπάθεια θα πρέπει να γίνει από την αρχή ουσιαστικά. Να δώσω όμω τώρα το λόγο στον κύριο Πολ Μέλη, ο οποίο είναι συμπατριώτης μου και είναι associate fellow του προγράμματο τη Αφρική του Chatham House. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σα πω ε, ευθύ εξ αρχή ότι πρόκειται για ένα ανεξάρτητο Έδρυμα ε, Εξέταση τη Εξωτερική ε, Πολιτική. Οπότε δεν παρουσιάζουμε εδώ τι προοπτικέ τη Βρετανική κυβέρνηση, αλλά αντιθέτω την δική μου προσωπική άποψη εγώ θα σα προβάλλω εδώ. Ε, δεν το πιστεύαμε, λέει και ο Πρόεδρο, έτσι καλώ. Ε, το Σαχέλ λοιπόν αποτελεί έναν ένα δύσκολο τομέα άσκησης εξωτερικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα ήθελα να σχολιάσω ε, λίγο και να συμπληρώσω τα όσα μας είπε μόλις τώρα ο κύριος Ελοζάντα ως προς το πώς διαμορφώνεται η περιοχή Σαχέλ και ποιες είναι οι προκλήσεις για την παροχή υποστήριξη από τη δική μας πλευρά ποιε είναι δηλαδή οι τη της ε, και θα σα δώσω κάποιε πρακτικέ λεπτομέρειε από την ίδια την περιοχή. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ένα-δύο πράγματα που είναι πολύ ε, προφανή και τα οποία ήδη ε, βέβαια εξέφρασαν, εξέφρασε ο κ. Σαλό. Η ανάπτυξη λοιπόν και η σταθερότητα και η ασφάλεια του Σαχέλ θα πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την ίδια την περιοχή, αλλά θα πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η αποτελεί το Σαχέλ μια πολύ κοντινή γειτονική περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μία από τις φτωχότερε περιοχές του κόσμου ε, και από τότε που υπάρχουν δείκτες κοινωνικής ανάπτυξης ε, έκτοτε είναι πάντοτε μία από τις στοχότερες ε, περιοχές, ενώ αντιμετωπίσει τώρα συμπληρωματικές ε, προκλήσεις όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η αύξηση του πληθυσμού η οποία έχει επιταθεί ακόμα περισσότερο κατά τελευταία χρόνια και βέβαια τώρα η τζιχαντιστική τρομοκρατία. Και βέβαια αυτά τα προβλήματα στην περιοχή έχουν αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει οξύ, οξία έλλειψη ε, βιώσιμων οικονομικών δυνατοτήτων ε, για τον ε, πληθυσμό, τον αυξανόμενο πληθυσμό του Σαχέλ με αποτέλεσμα να αυξάνεται η μετανάστευση προς την Ευρώπη. συχνά δηλαδή όταν κανείς ταξιδεύει άτυπα σε αυτή την περιοχή συχνά η ερώτηση που ακούει είναι πώς μπορώ να λάβω μια θεώρηση βίζα δηλαδή για να έρθω στην Ευρώπη και είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Ε, αν δεν υπάρχουν λοιπόν βιώσιμες δυνατότητες εκεί που μένει κανείς είναι προφανές ότι θέλουν να καταλήψουν. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ποια είναι η κινητήρια δύναμη, αν θέλετε, για αυτού του ανθρώπου. Επειδή δεν έχουν τι δυνατότητε να ζήσουν εκεί, προσπαθούν να βρουν πού αλλού μπορούν να βρουν τη δυνατότητα για τα προ το ζήν. Αυτέ λοιπόν είναι επιπτώσει σε επίπεδο μετανάστευση, σε πράγμα το οποίο βέβαια ε, καθιστά και πολύ σημαντική την περιοχή του Σαχέλ, ε, σημαντικό ζήτημα στο σχέδιο του, του σχετικού θεματολογίου. Αλλά ταυτόχρονα ε, και η τζιχαντιστική τρομοκρατία ε, σε, αυτόν τον, ε, σε αυτή την ευρύτερη περιοχή δεν απειλεί μόνο τη σταθερότητα των σχετικών ε, κρατών αλλά και των κρατών του Μακρέν, αποτελεί απειλή για την ευρύτερη δυτικοαφρικανική περιοχή. Και η Δυτική Αφρική ως συνολική περιοχή είναι βέβαια ε, μια περιοχή στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει τεράστιους πόρους ε, και επενδυτικά και σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας κατά τα τελευταία 20-30 χρόνια. Ε, και από τα μέσα του 1990 η εν λόγω περιοχή έχει καταδείξει σταθερή οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση των σχετικών κοινωνικών δικτών και αυξάνεται και ο εγγραμματισμός σε όλες αυτές τις περιοχές. Υπάρχει και η βελτίωση μέσω του ΕΚΟΓΟΣ και μόνο ένα κράτο υπάρχει, αν όχι ένα το οποίο δεν είναι καθόλου δημοκρατικό και μία-δύο ακόμα χώρες οι οποίες έχουν δημοκρατικά πολιτεύματα τα οποία δεν είναι πολύ σταθερά. Οι περισσότερες λοιπόν ε, χώρες ε, του Σαχέλ μπορούν πράγματι να επηρεάσουν τις κυβερνήσεις τους μέσω της κάλπης, ε, μέσω των μέσω ενημέρωση και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος σε αυτό το επίπεδο. Και το τι, το τι συμβαίνει λοιπόν στην περιοχή του Σαχέλ έχει αντίκτυπο στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αφρική. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους η Δυτική Αφρική και η περιοχή του Σαχέλ έχουν πάρα πολύ στενούς θεσμούς είναι η οικονομική τους δεσμή αλλά και η κοινωνική και εθνοτική δεσμή. Ε, για παράδειγμα, ε, ο πληθυσμός Χάουζα της Βόρειας Νιγηρίας αλλά και του κεντρικού και νότιου Μαλή είναι ουσιαστικά η ίδια εθνωτική ομάδα και απλώ του χωρίζει ένα σύνολο Και τέτοιου είδου κοινοί εθνοτικοί πληθυσμοί υπάρχουν και σε άλλε περιοχέ. Όταν βρίσκεται κανεί, για παράδειγμα, στην Βόρεια Νιγηρία, να βρίσκεται κανεί στο Νιαμέ, ε, βρίσκεται, συμμετέχει σε συναντήσει όπου ομιλείται η Χάουζα. Και ακριβώ, όχι τα γαλλικά. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η αίσθηση σε εκείνε τι ε, περιοχέ κοινή, αν θέλετε, κοινότητε. Ε, αλλά πέρα αυτών ε, θα πρέπει να πούμε ότι συχνά υπάρχουν τέτοιου είδους ε, κοινέ ε, κοινότητε, οι οποίες βέβαια δεν προσαρμόζονται στα σύνορα που άφησε αν θέλετε η περιοχή των Ευρωπαίων Και από εκεί και μετά υπάρχει για παράδειγμα, στη Νίγηρα υπάρχει μια εβδομαδιαία αγορά ζωικού κεφαλαίου ε, και από, είχαμε κάποιου εμπόρους από την Ιγυρία, από το Λάγος, οι οποίοι σε κάθε εβδομαδιαία τέτοια αγορά ε, μετέβαιναν στις παράκτητες αγορέ για να ε, τα πουλήσουν και επέστρεφαν στη συνέχεια. Δηλαδή έχουμε εμπορεύματα τα οποία ξεκινούν από τις ακτές των δυτικοαφρικανικών κρατών και αντίστοιχες, ε, ε, αντίστοιχα εμπορεύματα που έρχονται από τις ε, χώρες του Σαχέλ, αλλά και εργατικό δυναμικό, γιατί υπάρχει τέτοια έλλειψη. Και βέβαια, όπως ανέφερε ήδη ο κύριος Σαλόνζο, συχνά είναι περιφερειακό το φαινόμενο της μετανάστευσης στην ίδια την Αφρική. Δηλαδή συχνά από αυτές τις χώρες του Σαχέλ μετακινούνται προς τις παράκτιες χώρες του ώστε να εργαστούν εκεί στις σχετικές καλλιέργειες. Άρα λοιπόν, η Λύσει ε, που θα βρούμε θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητε της περιοχής του Σαχέλ και θα υποφεληθούν αν υπάρχει μια βιώσιμη στρατηγική που θα καλύπτει το σύνολο της Δυτικής Αφρικής και όχι μόνο του Σαχέλ. Και αν ρίξουμε μια ματιά εδώ στην, ε, στο, στο χάρτη, θα δούμε ποια είναι αυτή η γεωγραφική ε, πραγματικότητα. Αν δούμε δηλαδή από, τη, από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα δούμε ότι είναι πραγματικά τεράστια αυτή η ζώνη του Σαχέλ που περιλαμβάνει χιλιάδες χιλιόμετρα. Αν δούμε από το βορρά προς τον νότο τι συμβαίνει θα δούμε πως υπάρχουν ε, μία σειρά από οικονομικούς δεσμούς, για παράδειγμα Μαυριτανία και Σενεγάλη, ε, Μαλή και ακτή του Ελεφαντεστού, Μπουρκίνα Φάσο και Γκάνα, σε την Νιγηρία και Οπότε πολύ ε, ε, στενή οικονομική δεσμή αλλά και κοινά ε, έργα σε επίπεδο υποδομής που αναπτύσσονται και προωθούνται αυτή την περίοδο. Και κυρίως βέβαια οι χώρες τους Σαχέλ χρησιμοποιούν και το ίδιο νόμισμα, το φράγκο CFA. Το ίδιο δηλαδή νόμισμα το οποίο χρησιμοποιούν περισσότερες χώρες της γαλλόφωνης Δυτικής Αφρικής. Άρα λοιπόν υπάρχει εδώ κοινό θέλετε, μακροοικονομικό και δημοσιονομικό και επίπεδο πολιτική πολιτικής ε, πλαίσιο. Υπάρχει δηλαδή, υπάρχουν κάποια βασικά, αν θέλετε, σημεία, κοινά σημεία αναφορά σε επίπεδο μακροοικονομικής ε, πολιτικής ε, παρά το ότι έχουμε να κάνουμε διαφορετικές ε, χώρες. Για παράδειγμα η Κεντρική Τράπεζα στο Ντακάρ της Σενεγάλης είναι αρμόδια για το νόμισμα στο οποίο συμμετέχουν και άλλες χώρες όπως το Μαλί και ο Νίγηρας. Και από εκεί και μετά υπάρχουν και μία από σε μια σειρά από περαιτέρω περιφερειακά θεσμικά όργανα πέραν του Σαχέλ. Βέβαια, ο κ. Σανούς αναφέρθηκε στις ε, χώρες του G5, αλλά θα πρέπει να αναφέρουμε και το CLISS, ε, δηλαδή την ε, Περιφερειακή Ένωση που διοργανώνει αγροτικές δράσεις, δράσεις αγροτικές πολιτικές και όλες τις άλλες πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της ξηρασίας στην περιοχή θα ήθελα να μας υπερθυμίσω σε όλους μας ε, το γιατί είναι τόσο σημαντική η περιοχή του Σαχέλ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται στα νότια, θέλετε, στα νότια άκρα της Σαχάρας, αλλά ε, σχετίζεται η σημασία της περιοχής του Σαχέλ και με τον κύκλο της αγροτικής παραγωγής τροφίμων. Υπάρχει μόνο μία ετήσια εποχή των ε, βροχών από, τις, ε, από τα τέλη του Ιουνίου, αρχές Ιουλίου μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να παραχθούν οι περισσότερες, ε, για περισσότερα τρόφιμα, δηλαδή τα κυρία Δημητριακά. Ε, δημητριακά, ε, ίσως με κάποια ε, προσθήκη από κάποια ε, λαχανικά και ίσως με κάποια προσθήκη κρέατος ή ψαριού. Ε, και από εκεί και μετά υπάρχουν και κάποιες ε, εξαγωγικές ε, καλλιέργειες, για παράδειγμα όπως τα ΙΚΑΠΗ καριτέ, άλλοι. Και υπάρχει από εκεί και μετά, σε αυτή την περίοδο των βροχών έχουμε και την ανάπτυξη της χλωρίδας για την πόστιση των κοπαδιών. Από εκεί και μετά υπάρχουν κάποιες πηγές, κάποιες τοπικές λίμνες για την τήρηση κάποιων λαχανοκήπων, μικρής έκτασης καλλιεργείων λαχανικών και έχουμε και τα ε, αυτούς τους καρπούς, αλλά και τα δέντρα μάγκο τα οποία καλλιεργούνται. Όμως υπάρχει μικρό χρονικό αν θέλετε παράθυρο για όλες αυτές τις καλλιέργειες, πράγμα το οποίο εκθέτει την περιοχή του Σαχέλ, όχι μόνο στις αιτήσει ξηρασίες, οι οποίες, δηλαδή μια ξηρασία η οποία συμβαίνει ανά τρία-τέσσερα χρόνια. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο λαμβάνει χώρα ανατακτά χρονικά διαστήματα σε όλες τις χώρες του Σαχέλ ανά δύο ή τρία τέσσερα χρόνια, αλλά από εκεί και μετά πρέπει να ε, ληφθούν υπόψη τα ζητήματα και της ε, κλιματικής αλλαγής, αλλά και ε, ζητήματα ασφαλείας τροφίμων. Ένας από τους λόγους που η κρίση στο Μάλι ήταν τόσο σημαντική ήταν ακριβώς επειδή η κρίση είχε αντίκτυπο στην παραγωγή των αγροτικών τροφίμων. το 2012, δηλαδή μια περίοδο που βρισκόταν υπό την από τον έλεγχο των τζιχαντιστών είναι λόγω περιοχή. Άρα δεν ήταν δυνατό λοιπόν να, παρα, να παρασχεθούν σχετικές υπηρεσίες. Υπήρξε εκτοπισμός των ανθρώπων εκεί και κατά συνέπεια και μείωση της παραγωγής ε, και έλλειψη τροφίμων. Αλλά από εκεί και μετά η περιοχή έχει και κάποια ισχυρά στοιχεία και δεν θα πρέπει να τα υποτιμούμε. Και εδώ αναφέρομαι ιδιαίτερα στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. Από τη δεκαετία του 70 και του 80 όπου σημειώθηκαν πραγματικά ιδιαίτερα καταστροφικές εξηρασίες, οι χώρες του Σαχέλ ε, ένιωσαν ιδιαίτερα έντονα αυτές τις κρίσεις ε, και μάλιστα ήταν ε, πιο επίπονες από ό,τι οι πιο πρόσφατες κρίσεις. Μίλαγα με κάποιον στην Πουρκίνα Φάσο το Μάρτιο και μου είχε, πει ότι από την βορειότερη πόλη της Μπουρκίνα Φάσο στο Μάρτιο. Ε, ουσιαστικά όλος ο δρόμος ήταν διάσπαρτος από νεκρά ζώα. Ε, ήταν τόσο μεγάλη δηλαδή η έκταση της, ε, της κρίσης τότε την δεκαετία του 80. Δηλαδή προφανώς και τώρα είναι ιδιαίτερα καταστροφικές και οξύς οι κρίσεις, αλλά πραγματικά με σύγκριση εκείνες της κρίσης πριν από 40 και 50 χρόνια ήταν ακόμη χειρότερο και έκτοτε έχουν δημιουργήσει ένα πραγματικά εξαιρετικά εκτενές σύστημα παρακολούθησης, παρακολούθησης ε, των ε, καιρικών ε, συνθήκων και του ζωικού κεφαλαίου και της νοκαλλιεργιών. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί ακόμα και αν βρίσκεται κανείς σε μια απομενωμένη γωνιά της χώρας θα λαμβάνει κάποια δεδομένα, δεδομένα αξιόπιστα όχι από την, ε, Παγκόσμια Τράπεζα, οποιοδήποτε άλλο διεθνή φορέα, όχι από, την, από τις ίδιες τις ε, αρμόδιες αρχές όπου θα ε, λαμβάνουν δηλαδή πληροφορίες σε ό,τι αφορά το επίπεδο του υδροφόρου ορίζοντα, το ε, επίπεδο της αγροτικής παραγωγής τροφίμων και ό,τι καθεξής. Και υπάρχουν και συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα δύο-τρεις εβδομάδες ή και σε μηνιαίο επίπεδο στις επαρχίες αλλά και ετησίω σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων όλα τα σχετικά δεδομένα τυχάνουν επεξεργασία. Αρχικά λοιπόν αυτό το εργαλείο αναπτύχθηκε ούτω ώστε να αποφευχθεί η πλήρης καταστροφή γιατί το, τα διδάγματα που έλαβε κανείς από τις δεκαετίες του 70 και του 80 ήταν ότι αν δεν γνωρίζει κανείς το τι συμβαίνει θα υπάρξουν θάνατοι και ζώων και ε, θα χαθούν ανθρώπινες ζωές. Άρα λοιπόν από ένα τέτοιο εργαλείο για την αντιμετώπιση οξύων καταστροφών δημιουργήθηκε ένα εργαλείο το οποίο χρησιμεύει περισσότερο στην στο να καταστήσει την αγροτική παραγωγή πιο ανθεκτική. Με τη χρήση λοιπόν των νέων τεχνολογιών, smartphones και laptops, ηλεκτρονικών υπολογιστών και ούτω καθεξής, οι εν λόγω χώρες γίνονται όλο και πιο ισχυρές, δηλαδή πιο ικανές στην ανάλυση αυτών των δεδομένων, έτσι ώστε να γνωρίζουν ποιες είναι οι περιοχές στις οποίες ενδέχεται να σημειωθούν κρίσεις. Και Προφανώ υπάρχει εδώ μια προσπάθεια που πρέπει να γίνει σε εκπαιδευτικό επίπεδο, υπάρχει μια προετοιμασία που θα πρέπει να γίνει, αλλά τα πράγματα αλλάζουν, βελτιώνονται. Εγώ βρισκόμουν στο γραφείο ενό από του περιφερειακού διευθυντέ για την ε, ανάλυση ουσιαστικών δεδομένων πριν από κάποια χρόνια και χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν κάποιο ε, που βρισκόταν 1500 χιλιόμετρα ε, μακριά στα ανατολικά τη και ε, ήθελε να γνωρίζει πώς θα μπορούσε να τροφοδοτήσει κάποια δεδομένα μέσα στην, ε, στο σχετικό app, δηλαδή την εφαρμογή που είχε στο smartphone του. Δηλαδή ε, πράγματι η συλλογή αυτών των δεδομένων σε επίπεδο αγροτικής παραγωγής βελτιώνεται. Όμως κάτι άλλο που σημαίνει το εξή. Όλα αυτά γίνονται ή λαμβάνουν χώρο στο πλαίσιο ε, πολύ σημαντικών κοινωνικών αλλαγών. Και βέβαια η σημαντικότατη παράμετρος εδώ ε, είναι η αύξηση του πληθυσμού. Δηλαδή η αύξηση του πληθυσμού, το, ποσοστό αύξηση του πληθυσμού είναι από τα υψηλότερα ε, στον κόσμο. Στο Μαλέ για παράδειγμα, φτάνει το 3%, στον Νίγηρα το 4%, στην Πουρκίνα έφτασε το 2,1%. Όπω είπε και ο, ο αυτό σημαίνει ότι οι σχετικοί πληθυσμοί διπλασιάζονται εντό σε δύο δεκαετιών και στις ε, πόλεις των λόγω ε, χωρών ο πληθυσμός μπορεί να αυξάνεται ακόμα περισσότερο και αυτό βέβαια ασκεί τεράστιες πιέσεις στα σχετικά εδάφη, στους υδάτινους σπόρους αλλά και στην ικανότητα αυτών των ε, χωρών να παράσχουν στους πολίτες τους ένα βιώσιμο ε, εισόδημα. Υπάρχουν βέβαια λόγια να είμαστε αισιόδοξοι, δηλαδή οι κοινωνικοί δείκτες βελτιώνονται, υψηλότερο προσδόκιμο ζωής, ε, η εγγραφή στα σχολεία αυξάνεται. Όταν είχαν για παράδειγμα ανακοινωθεί οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας πριν από 15-16 χρόνια, ε, για τις περισσότερες χώρες του Σαχέλ ήταν εντελώς εξωπραγματικοί, αλλά βλέπουμε πως προσεγγίζουν, για παράδειγμα, το 30 5% των γυναικών και κοριτσιών στο Μαλί μεταξύ 15 και 24 ετών ε, είναι εγγράμματες και το 22% των ε, ε, ε, στην Μπουρκίνα Φάσο παρακολουθεί μια εκπαίδευση, ενώ το 69% των αγοριών και το 58% των κοριτσιών στον Νίκηρα ε, λαμβάνει πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή το δημοτικό. Και υπάρχουν και οι υποδομέ οι οποίε βελτιώνονται, κυρίω στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, αλλά και τα οδικά δίκτυα τα οποία είχαν. Ε, δεν είχα λάβει καμία προσοχή για δεκαετίες ε, να αναπτύσσονται. Για παράδειγμα, οι Κινέζοι ε, δημιουργούν ε, οδικά, οδικό δίκτυο, για παράδειγμα, στα νότια της Μπενίν για να τη συνδέσουν με τον Ήγηρα και την Πουρκίνα Φάσο. Και το Σαχέλ υποφελείται από την εγκύτητά του ε, με τη Δυτική Αφρική, αφού η Δυτική Αφρική αποτελεί μια από τι πιο ανθεκτικέ ε, περιοχέ στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Για παράδειγμα, με τι συνεργασία τη ε, ECOWAS και το κοινό δάσμολόγιο θα έχουμε ακόμα περισσότερη διευκόλυνση. Δηλαδή θα υπάρχουν σταθμοί συνολική διελευση μια στάση για την απλούστευση των σχετικών διαδικασιών και διασαφήσεων, αλλά βέβαια παραμένουν σημαντικότατε προκλήσει, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Για παράδειγμα, στον Ήγηρα μόνο το 29% λαμβάνει λαμβάνει η χώρα με την παρουσία δικαιωμένου προσωπικού. Μόνο το 21% των τοχετών. Στο Μάλι, μόνο το 11% των γυναικών μεταξύ 15 και 49 ετών χρησιμοποιούν μια σύγχρονη ε, μια σύγχρονη μέθοδο αντισύλληψης, ενώ στη Μαυριτανία από τις 100.000 ε, γεννήσεις ε, ζώντων νεοχρών, 602 μητέρε χάνουν τη ζωή του. Ε, στην Μπουρκίνα Φάσο ε, το ποσοστό του υποσυντισμού φτάνει το 30, ε, έφτασε το 31,5% το 2013, ενώ στο Νίγηρα έφτασε το 14,8% το 2014. Ε, βέβαια το τι ακριβώς είναι ένδια είναι λίγο αλλά με βάση τον ορισμό της Παγκόσμιας Τράπεζα το 53% του πληθυσμού του Μάλι ζει ακριβώς σε συνδικέ ένδιας, σε συνδίκες φτώχειας. Άρα λοιπόν η, βιωσιμότητα του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου των ε, χωρών του Σαχέλ είναι, ε, βρίσκεται υπό πολύ μεγάλη ε, πίεση και αυτό βέβαια οφείλεται στα όσα συμβαίνουν και με την κλιματική αλλαγή και παρά την εμπειρία που έχουν αυτοί οι πληθυσμοί στο να επιβιώνουν με περιορισμένους πόρους. Δηλαδή ε, υπήρχαν όλα αυτά τα προβλήματα προτού αρχίσει να λαμβάνει η χώρα η κλιματική αλλαγή. Οι ίδιες λοιπόν τώρα κοινωνίες ε, καλούνται να αντιμετωπίσουν και περισσότερες ε, προκλήσεις όπως η αποστεθαθερωτική βία και εγκληματικότητα. Έχουμε για παράδειγμα τις ε, κατά τόπους ε, εξεγέρσεις όπως τον του Αρέγ ε, στις περιοχές της Σαχάρα παραμένουν. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες εξεγέρσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει στο Μάλι που χρονολογούνται ήδη από τότε που απέκτησε η χώρα την ανεξαρτησία της και υπάρχουν ακόμα εντάσεις που παραμένουν μεταξύ εθνοτικών και κοινωνικών ομάδων καθώς μιλάμε συχνά για ιεραρχικού χαρακτήρα κοινωνίες. Έχουμε διενέξεις για παράδειγμα μεταξύ ε, αγροτών, ε, δηλαδή καλλιεργητών ε, της γης και ανεβηγών ζωικού κεφαλαίου κτηνοτρόφων για την χρήση των γεών. Αλλά όλες αυτές οι διαμάχες υπήρχαν ήδη από το παρελθόν, ενώ τώρα έχουμε να κάνουμε με την τρομοκρατία των τζιχαδιστών που διέπεται κυρίως από απολυταρχικού χαρακτήρα προσεγγίσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι ανοιχτή ε, σε διαμεσολαβήσεις. Ε, και από εκεί και μετά η εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών σε ολόκληρη τη Σαχάρα ε, δημιουργεί, εξασφαλίζει πολύ υψηλότερα έσοδα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά λαθρεμπόρια όπως παράδειγμα των ε, τσιγάρων, των τροφίμων, των ινοδοματοδών και ούτω καθεξής. Και βέβαια η αστάθεια εντείνεται ακόμα περισσότερο ακριβώ λόγω της διαμάχης μεταξύ των εκλογικών ομάδων για την έλεγχο αυτών των δρομολογίων. Και Γι' αυτό ε, χρειάστηκε τόσο πολλή χρόνο για την εφαρμογή τη Ειρηνευτική Συμφωνία ε, του Μάλι. Ε, δηλαδή, δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με ζήτημα εδώ επίλυση σε, πολιτικό επίπεδο. Έχουμε να κάνουμε και με τέτοιου είδου συμφέροντα εγκληματικών ομάδων. Από εκεί και μετά η κατάρρευση του καθεστώτο του Καντάφη στην Λιβύη απελευθέρωσε τεράστιε ποσότητε όπλων στη Σαχάρα. Σύγχρονων όπλων. Και μία από τις αιτίε που θεωρούνται, δεν είναι σίγουρο, ότι έχει οδηγήσει ακριβώς την αύξηση της βίας σε ό,τι αφορά την, ε, ε, το, το μαλλί ειδικότερα, είναι το γεγονός ότι οι δράσεις και των ε, γαλλικών δυνάμεων έχουν αρχίσει να Ακριβώ να περιορίζουν την τροφοδοσία αυτών των ομάδων με όπλα από την ε, Νότια Λιβύη. Οπότε οι σχετικέ ομάδε ε, προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα όπλα του από αλλού και γι' αυτό υπάρχουν τέτοιου είδους απεθέσει. Για παράδειγμα στο Δυτικό Νίγηρα έγινε μια τέτοια επίθεση σε ένα καταβλισμό. Δηλαδή είχαμε μια τέτοια ομάδα που ήρθε από το Μάλι και ε, η οποία σκότωσε 22 μέλη της, ε, των δυνάμεων ασφαλείας. δηλαδή δεν ε, άγγιξαν τους πρόσφυγες ή τα, τους ε, δικούς τους πόρους απλά έβαλαν φωτιά σε ένα στενοφόρο και από και μετά σκότωσαν όλους τους στρατιώτες ε, και πήραν τα όπλα τους. Και βέβαια, η, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών αλλά και η με την καταβολή λίτρων τους δίνουν ακόμα ε, περισσότερη δύναμη και βέβαια αυτές, αυτή του η δράση αποσταθεροποιεί ακόμα περισσότερο τις ε, χώρες του Σαγγέλ, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα του να παράσχουν και ε, ένα βιώσιμο τρόπο διαβίωσης στους ε, νέους τους. Για παράδειγμα, πώς μπορεί κανείς να βγάλει τα προστοζήν σε μια χώρα του Σαχέλ ως βοσκός. Ενώ αντιθέτω, εάν για παράδειγμα οδηγεί πικάπ, δηλαδή ένα αγροτικό με ανοιχτή καρότσα για του λαθρεμπόρου ναρκωτικών, χρειαστεί να μεταβεί μόνο δύο-τρει φορέ από το Νίγηρα στην Αίγυπτο και να επιστρέψει και από εκεί και μετά μπορεί να κρατήσει αυτό το ε, όχημα ε, για τον εαυτό του ως δώρο, δηλαδή 15.000 δολάρια όχημα. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσό το οποίο θα χρειαζόταν χρόνια για να βγάλουμε ένα έντιμο επάγγελμα. Υπάρχουν αυτά τα, αυτές λοιπόν οι τεράστιες προκλήσεις και ε, οι χώρε του Σαχέλ είναι στην πλειοψηφία του συνταγματικέ και δημοκρατικά πολιτεύματα, αλλά δεν έχουν του ε, κατάλληλου πόρου. Ε, και εδώ εκπρόσωπο ε, μίλησε σε ό,τι αφορά, αναφέρθηκε στο γεγονό ότι χρειάστηκε να μεταφερθούν πόροι από το πρόγραμμα των τριών ΕΝ, ούτω ώστε να ενισχυθούν οι στρατιωτικέ δυνάμει, οι ένοπλε δυνάμει. Γιατί ο Νίγηρα συμμετέχει και στην διακρατική ομάδα για την μετώπιση της ε, Μπόκο Χαράμ στην ε, Βόρεια ε, Νιγηρία και να μειωθούν οι επιθέσεις. Από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζει επιθέσεις από τρομοκράτες του Μάλι που επιτίθεται σε, σε καταβλισμούς στα δυτικά της χώρας και μετά έχει προβλήματα στα βόρεια όπου προσπαθεί να σταματήσει το λαθρεμπόριο όπλων από την Νότια Λιβύη μέσω του Βόρειου Νίγηρα προς το Βόρειο Μαλί. Και εδώ βέβαια συνεργάζεται με τις χαλικές ενοπλές δυνάμεις. Και από εκεί και μετά υπάρχει και το ζήτημα του τι θα πρέπει να γίνει με μεταναστευτικές ροές που περνάνε μέσα από το Αγκαντές. Και αυτό συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα. Δηλαδή ε, κάποιοι έχουν πει ότι ε, οι ένοπλες δυνάμεις ε, του Μάλιχ βοηθούν ουσιαστικά τε, τους διακινητές όμως ε, πραγματικά οι, τα λόγω αυτά δίκτυα είναι πραγματικά δεν έχουν καθόλου εδώ και απλά θα πέταγαν τους ανθρώπους στην έρημο αν δηλαδή δεν είχαν τους ε, κατάλληλα τρόφιμα και νερό. Και έτσι και συνέβη. Άρα το ΜΑΛ έχει να αντιμετωπίσει αυτή την τόσο πολύπλοκη διαδικασία ειρήνευση και επίση υπάρχει πρόβλημα στην πυκνοκατοικημένη περιοχή του Μόπτικ και είναι γεωρική αυτή η περιοχή, βρίσκεται στην καρδιά τη ε, ενδοχώρας και εκεί υπάρχει έξαρση βία και υπάρχει και επίση ε, δράση τη ε, Τζιχάντ που στρατολογούν και κάποιες άλλες τοπικές ομάδες όπως η Αμαντού και εκεί υπάρχουν επίσης προβλήματα σε σχέση με τα βοσκοτόπια, προστριβές και για κάποιο λόγο δεν λειτουργούν οι παραδοσιακές διαδικασίες επιλύσης αυτών των διαφορών. Οπότε και αυτό είναι μια σημαντική απειλή για την ε, σταθερότητα της χώρας όπως και η κρίση στον ε, Βορρά. Τι να πούμε τώρα, ποια απειλή είναι μεγαλύτερη, ποια εγώ και κούρευτο, αλλά τέλος πάντων έχει πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις. Ακριβώς γιατί αυτό θίγει τη γεωρική παραγωγή, το, το, το βασικό κορμό της και τη βασική περιοχή που αναπτύσσεται αυτή η δραστηριότητα. Και οπότε γι' αυτό το λόγο και η, η παροχή των υπηρεσιών δεν ε, λειτουργεί, ε, οι κυβερνητικές υπηρεσίες, οπότε πάρα πολλοί, ακόμα και οι πιο φτωχοί, όσον αφορά την παιδεία, δηλαδή στρέφονται στην ιδιωτική παιδεία. Και ένας φίλο ε, φίλος μου πήρε τηλέφωνο χθες. Αυτός εργάζεται σε ένα εστιατόριο, αλλά μόλις πούλησε το ποδήλατό του για να πληρώσει για το σχολείο του γιού του, γιατί είναι ιδιωτικό, τα δημόσια σχολεία δεν αποδίδουν και οπότε και αυτό χτύπησε το ήδη χαμηλό του εισόδημα. Οπότε εκεί μπορεί κυρίως να βοηθήσει η Ευρώπη πέρα από τα τεχνοκρατικά ζητήματα, δηλαδή έχουμε την ε, καθαρή ενέργεια, την αλλαγή του κλίματος, την ασφαλεία, την ασφάλεια, τις άλλες πρωτοβουλίες κλπ. Είναι, είναι το πώ μπορεί να βοηθήσει τι δυνατότητε των χωρών αυτών να παράσχουν τις βασικές κρατικές υπηρεσίες, να λειτουργήσει δηλαδή το κράτος. Και έτσι οι κρατικέ ε, δομές και σε περιφερειακό και σε κρατικό επίπεδο και σε κοινοτικό ε, να λειτουργήσουν γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι δομές. Οπότε μη υπάρχουσαν, είναι πιο ευάλωτο το κράτος και δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Οι χώρες του Σαχέλ είναι από τις πιο φτωχές περιοχές στον κόσμο. Αλλά θεωρούν ότι η Ευρώπη είναι εταίρος τους και ότι μπορεί να διαδραματίσει κάποιον ρόλο. Ας πούμε έχουμε την ρήτρα 96 της Συμφωνίας Κοτονού για τα θέματα της, της ε, διακυβέρνησης και αυτό είναι κάτι εύχριστο και νομίζω ότι έχει βοηθήσει ιδίω στην Πουρκίνα Φάσο, στο Μάλι και στον Νίγηρα και όλες αυτές οι χώρες ε, τελευταία πενταετία της βλέπουμε ότι δεν έχουν βοηθήσει, απειλείται η δημοκρατία και πάντα η εταιρική σχέση με την Ευρώπη όμως μέσα σε όλα αυτά ήταν κάτι το χρήσιμο και από πολιτικής πλευράς και από πλευράς ανάπτυξης. Και τώρα είναι κατά κλείδι να ξαναπούμε πόσο σημαντικέ είναι οι περιφερειακέ πρωτοβουλίε. Γιατί και εμεί ε, είμαστε μια περιφερειακή ε, πλατφόρμα και θεσμό. Οπότε θα πρέπει να συνεργαστούμε με το G5, να συνεργαστούμε με το ECOAS και με το CNSS που εξίσου είναι τέτοιε περιφερειακέ δομέ. Πώ σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο κύριο Στάνο. Πολύ καλή η παρουσίασή σου και να αρχίσει η συζήτηση με τον υποφαινόμενο, διότι έχω τρεις ερωτήσεις να σου υποβάλλω. Πρώτα πρώτα αυτό το οποίο είπα όταν ε, έλαβα το λόγο, ότι είπαμε ότι με το που θα ε, οι ζηχαντιστές στο Ισλαμικό κράτο στη Συρία και από εκεί θα έρθουν προς τα δόκια, άρα θα πρέπει να τους σταματήσουμε, να έχουμε συνορικούς ελέγχους, να δούμε τι θα γίνει την ασφάλεια. Επίσης ε, κάπου ανέφερε πάρα πολύ σύντομα την ε, αλλαγή του κλίματος τι κίνδυνοι υπάρχουν μακροπρόθεσμα για το Σαχέλ. Επίσης, τι γίνεται με τις μεταστηφτικές πίεσεις. Επίσης, Κίνα. Αναφέρθηκε σύντομα και η χώρα αυτή. Αλλά τι γίνεται ε, τώρα. Γιατί τώρα ίσως είναι πιο απομονωμένη η Αμερική με τον πρόεδρο Τραμπ. Άρα ίσως υπάρχει έδαφος για συνεργασία με την Κίνα. Ε, ακούγαμε ότι η Κίνα παίζει παντού στην ε, Αφρική και για το περιβάλλον υπήρχε κάποια συνεργασία. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε όμως ακριβώς εάν έχουμε απόσταση της Αμερικής από αυτό το χώρο και κάτι άλλο έτσι εσωτερικό μας. Πώς το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να συνεχίσει να έχει επαφή με αυτή την υπόθεση, δηλαδή μετά τον Brexit, τι μπορεί να κάνει για την σταθεροποίηση του Σαχέλ, μπορούμε να συνεχίσουμε να εμπλεκόμεθα σε αυτά τα δύσκολα προγράμματα, σε αυτά τα ακριβά προγράμματα. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε εμπλεκόμενοι σε αυτή την πολυμερή προσπάθεια. Τώρα, όποιο συνέδρο θέλει μπορεί να λάβει το λόγο. Πρώτα πρώτα. Από το ΕΛΚΟ, ο κύριος Μιλιάν Μον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον πρέσβητο τον κύριο ε, λοσάδα και άρχισα βέβαια να έρθω, έχασα την αρχή, μου φάνηκε ενδιαφέρουσα, πολύπλοκη αυτή η παρουσία του κυρίου Αλλά επίσης, τι γίνεται με την ενευτική διαδικασία στο Μαλί, τι γίνεται με την υλοποίηση ε, της συμφωνίας του Αλγερίου. Λέτε ότι τα πράγματα προχωρούν αργά αλλά σταθερά όμως αυτή τη μεσολάβηση, η διεθνή, όλων αυτών τι γίνεται. Είπαμε ότι έχουμε το ΣΕΝΤΕΟ, έχουμε τα Ηνωμένα Έθνη, έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που εμπλέκονται και μετά έχουμε και την G5, έχουμε ένα σωρό οργανισμού α και η Αφρικανική Ένωση. Όλοι αυτοί λοιπόν οι διεθνεί οργανισμοί και θεσμοί έχουν εμπλεκεί σε αυτή τη διαμεσολάβηση. έχουμε το θέμα τώρα τη παρακολούθησης, τη εξέλιξη, τη υλοποίησης αυτή τη νευτική συμφωνία. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε συντονισμό, ενότητα δράσης, μια που εμπλέκονται όλοι αυτοί. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ο συνάδελφος ο Γερμανός από τους Σοσιαλδημοκράτες. Α, τρεις, τρεις έχουν χτίσει το λόγο, οπότε να ρωτήσετε όλοι μαζί, να απαντηθούν όλοι μαζί. Κύριος Λίτς, ευχαριστώ και τους δύο εγώ εκπροσωπώ την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για το θέμα του καταπιστευματικού ταμείου. Ε, αναφέρεται πόσο σημαντικό είναι αυτό και εργαλείο σταθερότητας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για δύο πράγματα. Ε, τώρα ζητάμε πολύ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ε, μέσα ασφαλείας που μπαίνουν... Ε, στο χώρο της ανάπτυξης. Θα μπορούσατε να επεκταθείτε λίγο σε αυτό. Και μετά όταν μιλάμε για το καταπίστευμα για την Αφρική, υποθέτω, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τι ποσοστό πηγαίνει στην ασφάλεια και τι πηγαίνει επιτόπου στην κατάσταση για να βοηθήσει ε, να καταπολεμηθούν ε, τα αίτια της μετανάστευσης. Είτε αυτά είναι ε, η ανεργία, είτε υποδομές κτλ. Έχω και εγώ την ίδια ερώτηση επίσης για την Κίνα. Διότι όπως είπατε είναι, παίζει πολύ εκεί και με έργα υποδομών που χρηματοδοτεί και άλλα. Πώς αξιολογείται και πώς προβλέπετε την εξωτερική πολιτική της Κίνας σε σύγκριση με τη δική μας. ένα τελευταίο για την κλιματική αλλαγή. Έχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτούς τους συζητούν εκεί. Είναι θέμα που απασχολεί τις χώρες Σαχέλ. Και υπάρχει και ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής που έχει να κάνει με το κλίμα. Μετά τη Συμφωνία των Παρισίων θα πρέπει να έχουμε και ένα πρόγραμμα κλιματικών επενδύσεων. Αυτό το σκέφτονται οι χώρες αυτές για την ενεργειακή τους ασφάλεια και ο Ας ελπίσουμε ότι οι Πολιτείες δεν θα αποσυρθούν από τη Συμφωνία των Παρισιών. Γιατί θα είμαστε χαμένοι στο διάστημα αλλιώ. Ο κ. Μπούχνερ από τους Πρασίνους είναι ο τελευταίος που θέλει να ρωτήσει. Παρακαλώ. Κύριε Μπούχνερ, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Έχω μια τελείως διαφορετική ερώτηση εγώ. Εδώ εμεί συζητούμε βέβαια για την περιοχή του Σαχέλ, αλλά σε καμία από τις συμβατικές αυτές περιφέρειες δεν συμπεριλαμβάνεται η Δυτική Σαχάρα. Ξέρω ότι γεωγραφικά δεν ανήκει εκεί, αλλά είναι μια περιφέρεια τελείως παραμελημένη, όπου ο βασικός κλάδος της οικονομίας ε, ε, και το πιο παραγωγικό κομμάτι είναι η μαροκινή κατοχή. Πάρα πολύ σκληρή και πάρα πολύ καταπιεστική και μοσταγή. Και το υπόλοιπο κομμάτι ε, το αγνοώνει πάντες. Ε, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το τομέα. Δεν θέλω να, να παραμείνει έτσι και παραμελημένος αυτός ο χώρος. Όταν έκανα την έκθεσή μου και έβαλα μέσα τη Δυτική Σαχάρα, όπως φαντάζεστε, ε, κυριάρχησε κατά 95% ε, στη συζήτηση και ε, τον καυγά. Και ξεχάσαμε το Σαχέλ. Δεν θέλω τώρα να το ξαναφέρουμε αν είναι στο Σαχέλ, αν δεν είναι και ποιες είναι οι μελλοντικέ ελπίδες για την ανεξαρτησία κτλ. Είναι ξεχωριστή συζήτηση από τη σημερινή που μας απασχολεί, που είναι το ίδιο το Σαχέλ. Εδώ Α, και ο κύριος Βέντα θέλει να μιλήσει, ναι. Παρακαλώ. Να σας τα πω ισπανικά, να με καταλάβετε. Απευθείας κύριε Πρέσβη, είπατε για την κοινή προσπάθειά σας με την κυρία Μογγερίνη και είπατε και για τις γειτνιάζουσες χώρες, αλλά το πρόβλημα που τώρα αναδύεται στο Νότιο Σουδάν, ποιο είναι, ότι αυτά τα στοιχεία τα οποία ελάβαμε, ε, και εγώ ως ε, Επιτροπή ανάπτυξη είναι η ανθρωπιστική βοήθεια, τα σχετικά με αυτήν Και έχουμε τώρα αυτού όλου του ε, πρόσφυγες πάνε στην Ουγγάντα και είναι πάνω από 250.000. Οι πρόσφυγες λέω. Και ακριβώς όπως είπε και ο Επίτροπο Τηλιανίδη, ενδεχομένως έχουμε μέχρι τα τέλη ε, τη χρονιάς ίσως μια κρίση ανθρωπιστική του ενό εκατομμυρίου προσφύγων. Τι λέτε. Μπάς και δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Γιατί Οπότε φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα και με τις άλλες γειτονιάζες χώρες και όχι μόνο με το Σαχέλ. Άρα η Ουγγάντα θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την υποδοχή όλων αυτών των προσφύγων. Επίση, έχουμε το European External Investment Plan της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορά τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα της ε, Ένωσης για κάποιες ΜΜΕ στην Αφρική που έχουν πρόβλημα όχι με τη μετανάστευση, αλλά γενικότερα με το πρόβλημα των χώρων της περιοχής, το οικονομικό. Δεν έχουμε ακόμα εξωτερική τράπεζα επενδυτική, αλλά ίσως, την αποκτήσουμε στο μέλλον, λέει ο κύριος Στάνο Δεν ξέρω τώρα, έκλεισε ο κατάλογος των ερωτών των. έχετε τώρα, ε, εξοχότατε, θέλετε το λόγο πρώτος. αυτές τις δύσκολες ερωτήσεις. Ναι, ναι, εύστοχες, εύστοχες. Πρώτα, πρώτα, πρόεδρε. Ναι, πρόκειται για αυθεντική επιλευρά των ε, τρομοκρατών. Έχουμε δομές εξελίξεις σε Συρία και Ιράκ και όπως είπατε να δούμε τι σχέση υπάρχει μεταξύ των εκεί εξελίξεων γιατί αυτοί μπορεί να φτάσουν εδώ ε, Ευρώπη, Λιβύη, Μποκοχαράμ στην Ιγυρία. Πέντε χρόνια υπηρέτησα στην Ιγυρία. Ξέρω τη χώρα και η Μπόκο εκεί. Παρά το ότι λένε ότι συντονίζονται με το Ισλαμικό κράτος είναι κυρίως εσωτερικής εθνικής εμβέλειας στην Ιγυρία. Εκεί ξεκίνησαν, εξελίχθηκαν, αλλά τέλος πάντων είναι τοπικό κυρίως φαινόμενο. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να δημιουργηθεί ένας άξονας από Συρία σε Νιγηρία και μέσω Ευρώπης. Για πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα, όπως είπαμε, είναι πρόβλημα τοπικό της Νιγηρίας. Επίσης έχουμε αυτό το τείχος του Μπου. είναι είναι μια φυλή στη νότια Λιβύη και στο βόρειο Τσάντ αλλά και στη βόρεια Νιγηρία, σε αυτή την περιοχή, η οποία είναι κάθετη κατά του Ισλαμικού κράτους. Βεβαίω και εκεί υπάρχουν τζιχαντιστές, αλλά κοντράρονται. Ποτέ δεν θα επέτρεπαν επομένως να δημιουργηθεί τέτοιος άξονα. Και ξέρετε ότι έχω υπηρετήσει και στην Λιβύη για λογαριασμό του Ισπανικού κράτους. Επομένω, γι' αυτό σα προτεραιότητα και πρέπει να το επιλύσουμε οπωσδήποτε είναι το, θέμα τη Λιβύη. Αλλιώ δεν μπορεί να υπάρξει οριστική λύση για το Σαχέλ ούτε για την μετανάστευση ούτε για τίποτα άλλο. Και όλοι οι γητικοί πράγματα στην περιοχή λένε ότι τι θα γίνει με έλεγχο συνόρων, τι θα γίνει με το, με το δουλεμπόριο, τι θα γίνει αν δεν μπορούμε να συνηθούμε ημέν με του δε, ένθεν και εκείθεν των συνόρων. Άρα θα πρέπει έτσι να βρεθεί μια λύση. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε το θέμα της Λιβύης, το πρόβλημα της Λιβύης. Και άρα ε, είπαμε ότι έχει μεγάλη σημασία η ομοιογένεια αυτών των χωρών και να δούμε πώς θα συσχετίσουμε τα επιμέρους ζητήματα για να βρούμε τη λύση στο πρόβλημα Κίνα. Ξέρουμε ότι οι Κινέζοι δρούν παντού στην Αφρική. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο είπατε ότι τώρα με την νέα Αμερικανική πολιτική που δεν ξέρουμε καν πώς θα είναι ακριβώς, τι θα συμβεί. Τι θα φύγουν οι Αμερικανοί, θα τους υποκαταστήσουν οι Κινέζοι. Δύσκολο αυτό. Γιατί η ανάπτυξη είναι κυρίως αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πολλές πλευρές. Είναι θέμα οικονομικό, θέμα επενδύσεων. Τέλος πάντων είναι όμως ε, βαρύνων εταίρος. Οι Κινέζοι είναι και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και συμμετέχουν όλο ένα και περισσότερο στην ευτική διαδικασία. Ε, για αυτό ε, δεν θα μπορούσε να την καταστήσει κανείς, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούμε. Και για το Ηνωμένο Βασίλειο καλύτερα να απαντήσει ο βρετανό ε, συνάδελφο. Τώρα για την ενευτική διαδικασία στο Μάλι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο βουλευτή ε, Μιγιάν για την ερώτηση, γιατί ακριβώς αυτό είναι το κλειδί και η καρδιά του τι συμβαίνει. Έχουμε ένα βασικό πρόβλημα στην ευτική διαδικασία. Ουσιαστικό. Αυτό που περιέγραψε ο βουλευτής, δηλαδή, είναι το πρόβλημα της του ενιαίου χαρακτήρα της διαμεσολάβησης. Είναι πάρα πολύ περίπλοκη η νευτική αυτή διαδικασία και πάρα πολύ διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη ξέρουμε. Το έχουν υπογράψει αυτό η κυβέρνηση του Μάλι, την Ευτική Συμφωνία. Η πλατφόρμα που είναι η ομάδα των αποσυστικών κινημάτων, το ΕΡΕΓ, οι οποίοι ε, ήταν υπέρ της κυβέρνησης, αν και τώρα τα αλλάζουν λίγο, και επίσης οι τζιχατιστέ των Τουαρέκ, που είναι και, και, και στους Τουαρέκ Και οι τρεις το έχουν ε, συνυπογράψει, τη συμφωνία αυτή. Και ο, ο καθηγητής μου, Ντεμοντών, υπέγραψε μαζί με την ΕΚΟΓΑΣ, μαζί με την Αφρικανική Ένωση και ε, την Ισλαμική Οργάνωση και τα μέλη του G5 όχι ως σύνολα με τις πέντε χώρες που συμμετέχουν στην Στρογγυλή Τράπεζα στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Συν την Αργελία, ε, την Αλγερία που πρωτοστατεί και ηγείται όλες αυτές τις υπόθεσεις, ε, είναι επικεφαλής η Αλγερία. Κάθε μήνα λοιπόν συνεδριάζει στο Μάλι αυτή η Επιτροπή Παρακολούθησης και το πρόβλημα είναι να επιτύχουμε αυτόν τον ενιαίο χαρακτήρα, αυτή την ενότητα. Εμεί αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην τελευταία συνεδρίαση, κατόπιν δικού μα αιτήματο, είδαμε τον Πρωθυπουργό, τον ίδιο, και ε, προωθήσαμε ένα από τα βασικά θέματα της ενευτικής διαδικασίας που είναι η εγκατάσταση των ε, μεταβατικών αρχών. Μπορεί να ακούσατε ότι ε, στις 20 Νοεμβρίου θα γίνουν περιφερειακές τοπικές εκλογές. Αλλά ε, συγκρούονται διάφορες ομάδες ε, ε, στο βορρά που θέλουν και δεν θέλουν και απευθύνονται σε εμά για τη διαμεσολάβηση και προς τους Αλγερινούς. Και είμαστε όμοιροι των θέσεών τους και προσπαθούν να μας διχάσουν. Γι' αυτό ένα από τα βασικά στοιχεία όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίζει και αποφασιστικό ρόλο και το κάνει είναι να είναι ενιαία η φωνή της διαμεσολάβησης. Αυτό θα πρέπει να το προωθούμε πάντα μαζί με άλλες αρχές, πάση θυσία. Παράδειγμα, πολύ πιο συλλογική προσέγγιση και πάλι αυτή η έννοια το να ενστερνιστούν την Ευτική Συμφωνία οι ίδιοι. Η Νευτική Συμφωνία είχε ένα πρόβλημα. Ουσιαστικά επευλήθη έξωθεν από εμά. Α το αναγνωρίσουμε αυτό. Δεν υπάρχει σχέδιο Β. Ούτε οι αντάρτε ούτε τα κινήματα το έχουν υιοθετήσει, το έχουν εστερνιστεί αυτό το θέμα. Εκεί θα πρέπει να εργαστούμε και πάλι υπό την ηγεσία της Αλγερίας, γιατί αυτοί ε, κυριαρχούν Υπάρχει μόνιμη επιτροπή που σα είπα που συνεδριάζει κάθε μήνα για την παρακολούθηση και τέσσερι υποεπιτροπές ε, για διάφορα θέματα επιμέρου Συμφιλίωση, ανάπτυξη, θεσμών κτλ. Εκεί συμπροεδρεύει κάθε φορά η Αλγερία με κάποια άλλη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπροεδρεύει ε, με την Αλγερία για την ανάπτυξη σε αυτή την υποεπιτροπή. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να ενισχύσουμε τον ενιαίο χαρακτήρα της διαμεσολάβησης. Η επόμενη ερώτηση από τη Γερμανία για το καταπιστευματικό ταμείο. Η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ ε, ενδιαφέρουσα και αυτή. Διότι αν δούμε πώς προέκυψε αυτό το ταμείο, πώς γεννήθηκε, στην αρχή ήταν για το Σαχέλ και τα προβλήματα της περιοχής εκεί. Και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ε, ότι η Ισπανία ήταν η πρώτη που υπέγραψε με τον Υπουργό Εξωτερικών, Δημαργάγιο. Και ακολούθησε η τρομακτική μεταναστευτική κρίση. Είδαμε ε, τι γινόταν με ε, τη θάλασσα να ξεβράζει πτώματα παιδιών. Ε, αφόρητες εικόνες για όλους μας. παραμονές της Βαλέτας λοιπόν γεννήθηκε αυτή η ιδέα για το καταπιστευματικό ταμείο και είχε έρθει η ώρα να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που ήταν πραγματικά ε, φοβερό και κινδύνευε να αταράξει η θέμελα την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρθε λοιπόν αυτό το καταπίστευμα για να καταπολεμήσει τις βαθιές αιτίες της μετανάστευσης. Όπως σας είπα, Και μετά προσθέθηκε και το κέρας της Αφρικής. Υπάρχουν λοιπόν δύο στοιχεία, Σαχέλ και κέρας Αφρικής για τη μετανάστευση. Και προσθέθηκε και ένα τρίτο στοιχείο που είναι η Βόρεια Αφρική, δεν έχει ακόμα ανοίξει αυτή η θηρίδα στο ταμείο. Άρα το καταπιστευματικό ταμείο λειτουργεί για την ανάπτυξη, ακριβώς για το περιφερειακό πρόγραμμα δράσης για το Σαχέλ. Στη συνέχεια αν θέλετε μεταξελίχθηκε, μεταλλάχθηκε για να αντιμετωπίσει τη μετανάστευση και τώρα η μετανάστευση έρχεται να συναντήσει την ανάπτυξη. Συνδέεται πάρα πολύ με το θέμα της ασφάλειας και της κατοχής του εδάφους, της επικράτειας. Όταν παρετείται το κράτος και δεν είναι παρόν σε μία επικράτεια, μπαίνουν τα διάφορα λαθρεμπόρια, διακινητές και η ε, τρομοκρατία που πάντα λαθρεμπόριο γινόταν στην περιοχή. Ε, η αναστάθ... Ε, ανασφάλεια λοιπόν, που επικρατούσε στο βόρειο Μαλί τώρα κατεβαίνει προς τον νότο και ε, απειλεί την ειρήνη σε όλη την περιοχή. Θα πρέπει λοιπόν το Ταμείο αυτό να αντιμετωπίσει και θέματα ασφαλείας που έχουν όμως άμεση ή έμεση σχέση με τη μετανάστευση. Με ρωτήσετε και για τα ποσά. 36 είναι τα έργα που εγκρίθηκαν ήδη, αν δεν απατώμε, 575 εκατομμύρια ε, είναι 60% από το 1,1 δις του συνολικού ποσού. Το Νοέμβριο λοιπόν τέλη του μηνός θα έχουμε και πάλι μια νέα ε, συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για να δούμε ε, ποια θα, νέα έργα θα εγκριθούν για τη μετανάστευση. Αλλά αυτό το στοιχείο της ασφάλειας παραμένει κυριαρχό και στο G5. Για την Κίνα. Νομίζω απάντησα για την κλιματική αλλαγή. Να απαντήσει τίποτα άλλο και ο συνάδελφός μου, να μην τα απαντήσω όλα εγώ. Τρίτο για τη Δυτική Σαχάρα, νομίζω ότι ο πρόεδρος απάντησε θαυμάσια. Α, από την άλλη, στην εντολή μου έχω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και αυτό είναι η σχέση Ευρώπης, Μαγκρέμπ, Σαχέλ. 5-5-5. Δηλαδή είναι το G5. Οι, οι πέντε χώρες του Μαγκρέπ είναι η Ευρώπη. Ε, πολύ σημαντικό στοιχείο. Κάνω διάφορα σεμινάρια και πρόκειται να έχουμε και άμεσες επαφές και σε υπουργικό επίπεδο και όσο γίνεται υψηλότερο επίπεδο για το πώς θα διαρθρώσουμε αυτό το διάλογο που είναι πάρα πολύ δύσκολο ακριβώς γιατί τσακώνονται συνέχεια το Μαρόκο με την Αλγερία. Το θέμα είναι πολύ περίπλοκο, είναι πολύ λεπτό και ευαίσθητο. Υπάρχει μια φοβερή κόντρα εκεί. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τις σχέσεις τους αλλά κυρίως να μην θίξουμε τη Δυτική Σαχάρα, δεν είναι στην εντολή μου, αλλά άμα ανοίξει αυτός ο ασκός του αιώλου, χαθήκαμε. Σφυγκοφολιά είναι. Κύριε Βέντα, με ρωτήσετε για τον Νότιο Σουδάν και αυτό είναι εκτός της εντολής μου. Μιλήσατε για τους πρόσφυγες. Ε, με Α, θα μιλήσω και ισπανικά, γιατί και εσείς ισπανικά ε, με ρωτήσατε και με χαρά να απαντήσω ε, στη μητρική μου. Αυτό το θέμα των προσφύγων δεν το συζητάμε συχνά σε σχέση με τα προηγούμενα. Δηλαδή, έχουμε μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση, όχι μόνο μεταναστευτική. Ε, στην περιοχή της Λίμνης ε, του Τσάτ, ο Νίγηρας αντιμετωπίζει τριπλή κρίση. Λιβύη, Μάλι και Μπόκο Χάραμ ε, το Τσάτ αντιμετωπίζει την κρίση της Κεντρικής Αφρικής, την κρίση του Σουδάν και κυρίως ε, τους έπιασαν και στα πράσα ε, η Μπόκο Χαράμ. Είναι ανθρωπιστική κρίση που θα έρθει μπροστά μας, πολύ προσεχώς. Από εμπορικής πλευράς υπήρξε μια πολύ σημαντική συναλλαγή Τσάντ Νιγηρία ε, γινόταν πολύ μεγάλο εμπόριο σε διάφορες ζωοπανηγύρεις που μετακινούσε πληθυσμούς, εκατομμύρια κυκλοφορούσαν και πουλούσαν τα ζώα τους. Και αυτό σταμάτησε απότομα και βία. Και η πολιτική κρίση και η τρομοκρατία που προκάλεσε τον Πόκο Χαράμ από την ομότητα και τη βιότητά το οδήγησε και σε ανασφάλεια ολόκληρη την περιοχή. Και το Τσάντ που είναι μια ε, χώρα πολεμοχαρής από γεννησιμιού της, υφίσταται ε, πραγματικά ε, τεράστια πίεση. Έχουμε μια πολυεθνική δύναμη, έχω συμμετάσχει, έχω πάει πολλές φορές, πέντε χώρες θέλουν να παίξουν εκεί ρόλο, ε, ε, αμυνόμενες της περιοχής μαζί με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει δώσει δάνειο 50 εκατομμύρια ευρώ μέσω του μέσου σταθερότητας 50 εκατομμύρια ευρώ δάνειο ε, έχουμε ένα ε, πρόβλημα ανθρωπιστικό πρώτης τάξεως που αργά ή γρήγορα θα σκάσει μπροστά μας και θα μας κατακλείσει. Αυτό αφορά το Σαχέλ. Για το Σουδάν σας είπα δεν είναι δική μου περιοχή. Υπάρχει άλλος ειδικό εκπρόσωπος. Ε, το τσάτ πάντως είναι εύθραυτο και προεδρεύει στην Αφρικανική Ένωση. Προεδρεύει στο G5 και προεδρεύει και στις πρωτοβουλίες για τις στρατηγικές του Σαχέλ. Είναι και η έδρα της επιχείρησης Μπαρκάν και της πολυεθνούς δύναμης και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είναι και η χώρα από όπου καταγέται ο αρχηγός της αποστολής Μινούσμα, ο Αναδίδ, που είναι ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας ε, όλης της Μινούσμα, της ε, επιχείρησης στο Μάλι. Το Τσάτ λοιπόν είναι μια χώρα ε, πάρα πολύ ε, κρίσιμη, πολύ σημαντική. Ε, πολεμάνε, δεν έχουν πρόβλημα, είναι πάρα πολύ θαραλέοι. Πολλές φορές είναι και πολύ ε, ρυψοκίνδυνοι και ξέρει και να αμήνεται, αλλά έχουν τεράστια ανθρωπιστική κρίση που επίκειται. Αυτά, Πρόεδρε, νομίζω απάντησα. Και σας ευχαριστώ όλους για τα ερωτήματά σας. Ναι, κύριε Πρέσβη, έχετε πραγματικά πολύ βαθιά γνώση αυτού του περίπλοκου ζητήματος ε, και γι' αυτό νομίζω πως ε, πραγματικά διαφαίνεται γιατί χρειάζεται να έχουμε ένα συντονισμό μεταξύ μας. Ε, πολύ δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσεις όλα αυτά τα ζητήματα και τις κλιματικές αλλαγές. Βέβαια δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσεις το ζήτημα του Brexit γιατί είναι πολιτικός ευαίσθητο. Ναι, σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. να πω ότι η ιδιαιτερότητα της ε, κρίσης της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τα όσα έχουν αντιμετωπίσει οι χώρες ε, του Σαχέλ ε, έγινε στο γεγονός ότι ενώ είχαν αναρτά χρονικά διαστήματα ξηρασίες σε αυτέ τι χώρε, ανά 2, 3, 4 χρόνια και κάποιε πλημμύρε, γιατί πλημμύρε λαμβάνουν χώρα ανά χρονικά διαστήματα αλλάζει η γεωγραφία του. Και στι παλαιότερε προκλήσει είναι συνηθισμένε να αντιμετωπίζουν τέτοιε προκλήσει αυτέ οι χώρε, αλλά όχι τι νέε. Για παράδειγμα, εάν μιλάμε για βοσκοτόπου παραδοσιακού οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να διατηρηθούν ω ε, ε, τέτοιου είδου βοσκότοποι, γιατί ερημώνονται όλο ένα και περισσότερο, είναι δύσκολο. Δηλαδή, οι επιμένες αυτοί που διέσχιζαν αυτές τις περιοχές ε, προς τα νότια, θα αρχίσουν να θέλουν να εγκαθίστανται πιο μόνιμα στα νότια και αυτό θα οδηγήσει σε, ε, και οδηγήσει σε εντάσεις με τους ανθρώπους οι οποίοι ήδη βρίσκονται εδρεωμένοι εκεί και έχουν αγροτική δραστηριότητα. Και θυμάμαι σε μια επαρχιακή πόλη στον Ήγυρα που μιλούσα με έναν κτηνοτρόφο και μου έλεγε πως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά του είναι το γεγονός ότι κάθε χρόνο οι αγρότες οι οποίοι καλλιεργούν συγκεκριμένες εκτάσεις ε, τώρα δέχονται αυτές θέλετε, τις επισκέψεις ε, των, ε, των επιμένων και αυτό που κάνουν είναι εκεί που οι αρμόδιοι από τις εθνικές αρχές οριοθετούσαν τις συγκεκριμένες περιοχές που προορίζονταν για τις καλλιέργειες αλλάζουν με τους ε, με όσου μετακινούνται ακριβώ για να βοηθήσουν στα κοπάδια, με αποτέλεσμα να αλλάζουν και οι σχετικέ οριοθετήσει, να μην ισχύουν δηλαδή αυτέ κάθε χρόνο. Ε, και ε, από εκεί και μετά υπάρχει και το ζήτημα τη λίμνη Τσάντ και συζητείται εδώ και καιρό κατά πόσο συρρυκνώνεται ή όχι αυτή η λίμνη. Και πρόκειται για ένα ζήτημα δηλαδή το οποίο δημιουργεί διαφορέ. και αντιθέσεις. Εάν πάντως σκεφτούμε ότι οι χώρες του Σαχέλ ήδη δέχονται πιέσεις από άποψη ε, αύξησης του πληθυσμού και από άποψη πολιτικής αστάθειας. Έχουμε τώρα και την τρομοκρατία και την κλιματική αλλαγή που έρχονται να προσθεθούν ως ε, προβλήματα. Και ε, η χλωρίδα προφανώ, δηλαδή και η βλάστηση, μπορεί να αντικατασταθεί μόνο με συγκεκριμένου ρυθμού, Αυτό που επιτρέπει η φύση. Δεν μπορεί δηλαδή να επιταθεί ε, η όλη αποκατάσταση. Και το σύστημα που έχει δημιουργηθεί κατά πολέμηση της εξηρασίας στο CILSS είναι μεν πολύ ανθεκτικό, αλλά από εκεί και μετά θέλουμε μια πιο στρατηγική σκέψη ως προς το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή σε επίπεδο Σαχέλ και σε επίπεδο Δυτικής Αφρικής. Μια τέτοια στρατηγική για αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα, αλλά θα πρέπει να μπει στην ημερήσια διάταξη για αυτή την περιοχή. Ειδικότερα αφού ε, ε, οι απόψεις από την πλευρά των ίδιων των χωρών δεν είναι τόσο ε, σαφείς. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση συνήθως έχει ε, πολύ συγκεκριμένε απόψει, οπότε θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα είδο τεχνική, αν θέλετε, εταιρική σχέση με τι χώρε του Σαχέλου, ώστε να εξεταστεί το πώ ακριβώ μπορούν να αντιμετωπίσουν από κοινού την κλιματική αλλαγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, την πρωτατική πολιτική. Νομίζω πως ο, ο κύριος ε, Τάνεκ έχει δίκιο σε αυτό που είπε, ότι δηλαδή θα είναι αδύνατο η Βρετανία να δημιουργήσει το δικό της ανεξάρτητο και ευρύτατο πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τις ε, χώρες του Σαχέλ. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό που κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο είναι να εργάζεται ή το αρμόδιο δηλαδή Υπουργείο Αναπτυξιακής Εργασία, μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων, Oxfam, χριστιανικές οργανώσεις και άλλες, οι οποίες πράγματι έχουν δράσει σε αυτές τις χώρες ε, του Σαχέλ, αλλά τέτοιου είδου μη κυβερνητικέ οργανώσεις δεν έχουν στρατηγικού ακριβώ επίπεδου δυνατότητε. Δηλαδή είναι πολύ καλέ σε ό,τι αφορά την ε, κατατόπου συνεργασία με τι επιμέρου κοινότητε και ούτω καθεξής, αλλά δεν μπορούν να, να, να, να χαράξουν στρατηγική αυτέ οι μη κυβερνητικέ οργανώσει για το σύνολο του Σαχέλ. λοιπόν ή ε, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο θα ολοκληρώσει τη διαδικασία εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να εδραιώσει μια εταιρική σχέση, η οποία ακριβώ θα θεσμοθετήσει, αν θέλετε, ένα σύστημα με την ε, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χάραξη πολιτικής ε, στο Σαχέλ. Ας πάρουμε για παράδειγμα την αποστολή εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων, την EUTM. Εκεί συμμετέχουν συχνά Βρετανοί προσωπικό από το Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτή την ε, εκπαίδευση και νομίζω πως αυτό το προσωπικό θα είναι σε θέση να συνεχίσει να προσφέρει αυτή την υποστήριξη ακόμα και όταν η, Ευρωπαϊκή, η Μεγάλη Βρετανία αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά χρειάζεται ένα γενικότερο στρατηγικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί αυτό. Νομίζω για παράδειγμα πως η Νορβηγία ήδη έχει συμμετάσχει σε εκτεταμένο βαθμό στην εκπαιδευτική αποστολή την UTM και στην αποστολή στην ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Και εκεί συμμετείχαν στην εν λόγω αποστολή και ε, ενόπλες δυνάμεις από την ε, Γεωργία. Οπότε υπάρχουν μία σειρά από τομείς στου οποίου μπορεί να συμμετάσχει. Είτε πρόκειται δηλαδή για αναπτυξιακή βοήθεια ως χρηματοδοτική δηλαδή υποστήριξη. Όταν για παράδειγμα παρέχει τέτοιου είδου ε, υποστήριξη, χρηματοδοτική δηλαδή, σε επίπεδο προπολογισμών αυτών των ε, χωρών, προφανώ αν θέλει να πράξει το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο θα ήταν πιο λογικό να μην το κάνει ανεξάρτητα, αλλά να το κάνει μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό, για παράδειγμα, γίνεται και μέσω τη ε, εκπροσώπηση άλλων ευρωπαϊκών χωρών μέσω των πρεσβειών συγκεκριμένων κρατών μελών. Για παράδειγμα, έχει στο Μάλι μια εκπροσώπηση, αλλά όχι στη Μαυριτανία, όχι στον Νίγηρα, ούτε στο Τσάντ, αν θυμάμαι καλά, ή εν κάποια διπλωματική αποστολή στο, στο Ναι, υπάρχει μια Βρετανική αντιπροσωπεία, δύο άτομα συγκεκριμένα, τα οποία όμως ε, εντάσσονται, αν θέλετε, στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα του. Άρα, ναι, θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε το τι θα κάνουμε. Δηλαδή, ναι, λέμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τι ε, χώρε του Σαχέλ και τη Δυτική Αφρική, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα, ε, συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες δεν έχει υπάρξει ε, ισχυρή παρουσία και ορατή παρουσία του Ηνωμένου Βασίλειου, οπότε εκεί θα χρειαστεί και υποστήριξη. Τώρα το πώς θα χαράξει τη δική της εξωτερική πολιτική ως χώρα είναι κάτι διαφορετικό, αλλά από εκεί και μετά οτιδήποτε αποφασιστεί από εκεί και μετά να γίνει ανεξάρτητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά ε, αποστολή ενόπλων δυνάμεων, υποστήριξη και ούτω καθεξής, ε, θα δημιουργήσει προβλήματα, θα δημιουργήσει τριβές δηλαδή, αν δεν υπάρχει συντονισμός με την ευρωπαϊκή πολιτική. Συγγνώμη που σας στριμώξαμε λίγο, αλλά ναι, έτσι, έτσι, θα, θα φουντώνει η συζήτηση στους αμέσως επόμενους μήνες και από δική σου πλευρά ενδιαφέρον να δούμε πώ είναι η Βρετανία να μείνει κοντά σε όλε αυτέ τι δομές τη επιτροπή Άμυνα, εξωτερική Πολιτική κλπ. κλπ. Οπότε θα κάνουμε και οικονομίε ε, ε, κλίμακα, να δούμε τι θα γίνει με τι διμερεί ε, επαφέ κλπ. Χρειάζεται χρηματοδότηση σε όλε αυτέ τι χώρε. Έτσι κι αλλιώ είναι συσήφιο σχεδόν το έργο που έχουμε κάνουμε εκεί πέρα. Και ακούσαμε πάρα πολλά εδώ από τους ειδικού που καλέσαμε. Πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα. Και με εκείνη την έκθεση ο ίδιο ε, πριν από τρία χρόνια είδα τι γίνεται, τι έγινε με το G5 και είδαμε ότι τώρα έχουμε προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα ε, εντελεχέ. παραμένει φυσικά ευάλωτη αυτή η περιοχή και επομένω αυτό θα είναι πρόβλημα, θα είναι πρόκληση για το προβλέψιμο μέλλον με του τζιχαντιστάς και θα, με, ε, αυτό που εγώ ονομάζω λεωφόρο της τρομοκρατίας από Σομαλία μέχρι το Σαχέλ ε, ε, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να τα αγνοήσουμε και θα μας απασχολήσουν επομένω στο άμεσο μέλλον. Σας ευχαριστώ έτσι αλλιώ, κύριοι για όσα μας είπατε να κάνουμε ένα μόνο λεπτό διάλειμμα και κατόπιν θα δώσω τη σκητάλη στον κύριο Κούκαν. Good afternoon, ladies and gentlemen. Now we shall take... Γεια σας κυρίες και κύριοι. Για να δούμε τώρα το θέμα μας υπαριθμών 5 που είναι αυτή η σύναψη της ε, οικονομικής και προεξημένης μεταξύ των Καναδάφινων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφετέρου. CETA, as you know, was adopted by the Council. Η ΣΕΤΑ βγήκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και προσυπογράφηκε στις, ε, το τον Οκτώβριο του 2016, αλλά πρώτα είχαμε διάφορα ε, δραματικές ε, εξελίξεις και ενστάσεις τελευταία στιγμή από τα Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η συμφωνία που ονομάζεται ΣΕΤΑ είναι πάρα πολύ εντελεχής, είναι νομικά δεσμευτική και αφορά 1598 σελίδες. Αποτελείται από τόσες σελίδες. και πρόκειται και κάποια ε, στρατηγική συνεργασία όσον αφορά τις σχέσεις μας με τον Καναδά. Χρειάζεται η σύμφωνη νομή του Κοινοβουλίου για να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Πρόκειται το ICS, Σύστημα Επενδύσεων. Και πρόκειται επίση και μια συμφωνία πρέπει να ακυρωθεί από τα κράτη-μέλη. Στην ντα πρόκειται να γνωμοδοτήσουμε γιατί η ντα είναι κυρίω αρμόδια επιτροπή. Και όσον αφορά αυτή τη συμφωνία τη στρατηγική εταιρική σχέση θα πρέπει να περιμένουμε επίση και την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου. Οπότε και η ΑΦΕΤ θα καταστεί μετά η κυρίω αρμόδια επιτροπή. Έχουμε συγκριτή τον Τσολθάνο ο οποίο και θα λάβει το λόγο για να μα κάνει τη σχετική εισήγηση. Ευχαριστώ πολύ, Έντορτ. Ε, ε, σαν ηθοποιός έτσι πολλά ρόλους. Από πρόεδρος έγινα εισηγητής μέσα σε πέντε λεπτά. Αυτές είναι μεταμορφώσεις. Πολύ σημαντική συμφωνία αυτή. Ε, σχεδόν ε, βήθησε σε μια κρίση την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ πρόσφατα όλο αυτό το θέμα της συμφωνίας ΣΕΤΑ με τα δικαιώματα περιφερειακών κοινοβουλίων. Είδατε τι έγινε με την Βουλή της ε, Βαλονία που κόντεψε να ανατρέψει μια επταετή σχεδόν διαπραγμάτευση. Ε, την ενδεκάτη ώρα λύθη το θέμα, ήμασταν όλοι με κομμένη την ανάσα, επιτέλους λύθηκε. Φαίνεται ότι διασκεδάστηκαν οι φόβοι και ανησυχίες. Ε, δεν είμαι απολύτως βέβαιος τι συμφώνησε ο Βέλγος Πρωθυπουργός με τη Βαλονική Βουλή. Θα βγουν κάποια στιγμή αυτά στη φόρα. Πάντως η συμφωνία είναι ε, γενική, σύγχρονη, 1598 σελίδες αν δεν απατώμε και στη χώρα μου εκείνοι που πιστεύουν ότι με το Brexit θα ε, επαναδιαπραγματευτούμε 60 συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών ε, εν μία νυχτή θα μπορούν να συνεχίσουν να ονειρεύονται. Είναι μακριά ανοιχτωμένοι. Είναι πάρα πολύ μακρά διαπραγμάτευση και έχουμε και επίμαχες ε, διατάξεις. Το SDS, ε, στο SDS, το σύστημα επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους, ε, που μάλλον έχει πεθάνει. Θα δούμε τι θα γίνει με τη νέα κυβέρνηση το Γενάρη στις ΗΠΑ. Ο Καναδάς δεν στο παραπέντε. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει μέλλον και η ναύτα, η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών για τη Βόρεια Αμερική. Ο κύριος Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θέλει να επαναδιαπραγματευτεί και αυτή τη συμφωνία. Γενικά είναι πάρα πολύ ασταθέ και αβέβαιο το παγκόσμιο κλίμα ως προς το εμπόριο και την εξωτερική πολιτική. Πάντως, εγώ είμαι κάτι ενθουσιασμένος που ξεπέρασε αυτή την εμπλοκή η ΣΕΤΑ που Προκάλεσε Βαλονία στο παραπέντε. Τώρα τα κράτη-μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια και οι κυβερνήσει έχουν τον τελευταίο λόγο και μετά ελπίζουμε να τεθεί σε προσωρινή ε, ισχύ, ε, δεν απατώμε, ε, του χρόνου ακόμα και πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσης από όλα τα κοινοβούλια κτλ. Όπως σας είπα, η γνωμοδότηση είναι σχετικά σύντομη βασικά δίνει τη σύμφωνη γνώμη της δικής μας Επιτροπής στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, ίντα, αρμόδια επί της ουσίας είναι αυτή. Ο Καναδάς είναι πάρα πολύ στενός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει πάρα πολύ όρημη δημοκρατία και οικονομία. Ελπίζω να κάνουμε εμπόριο σε διάφορους τομείς με ένα πολύ καλό τρόπο. Με περίεργη διάβασα στο Βρετανικό τύπο ότι προβλέπεται για την επόμενη διετία πριν έρθει το Brexit να υποφεληθεί κατά 20% αύξηση του διεθνούς εμπορίου με το διμερούς με τον Καναδά η Μεγάλη Βρετανία. Και θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο κρίμα για τη χώρα μου που έχει μοναδικές σχέσεις με τον Καναδά. Γιατί έχουμε και το απικιακό παρελθόν και το, την ε, πράξη Βρετανίας Βορείου Αμερικής που είναι ουσιαστικά το Σύνταγμα του Καναδά και είναι ένα κοινοβουλευτικό δικό μας νομοθέτημα. Ήταν κρίμα να φύγει η Βρετανία από όλες αυτές τις συμφωνίες και πρέπει να βρει έναν τρόπο να παραμείνει προσιλωμένη και συνδεδεμένη με αυτές. Γενικά λοιπόν είναι προς όφελός μας και ο Πρωθυπουργός Τρουντό και οι διαπραγματευτές όλοι είχαν έρθει στις Βρυξέλλες πρόσφατα και είχαν δυσαρεστηθεί γιατί νόμιζαν ότι θα ναυαγούσε η προσπάθεια αυτή στο παραπέντε. Όπως σας είπα όμως ελήθηκε ευτυχώς να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας. Ελπίζω να έρθουν και τροπολογίες. Πότε η προθεσμία αύριο, στις 15 Νοεμβρίου, αύριο το μεσημέρι στις 12. Ωραία. Θα δούμε αν θέλει κανείς να καταθέσει καμιά τροπολογία. Δεν μπορώ να φανταστώ να υπάρχει μεγάλη αντίρρηση από τις μεγάλες πολιτικές ομάδες επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, on behalf of EPP Group, I... Uh, ε, για το ΕΛΚ. Ο αντικαταστήτη κύριο Κόβετσεφ που είναι ο σκιώδης ηγητής. Θα μίλησω στη θέση του γιατί είχε ένα πρόβλημα ε, με το αεροπλάνο. Τέλος πάντων είχαμε αυτό το σχέδιο κειμένο. Και λέει ο κ. Κοβατσέφ ότι 100% συμφωνεί με το κείμενο του κυρίου Τάνοκ. Και όσον αφορά αυτή την σύντομη αιτιολόγηση, όπως επίσης και με την ε, σύσταση για να δοθεί το πράσινο φως ε, στη Συμφωνία ΣΕΤΑ που είναι η πιο σύγχρονη ε, συνθήκη που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με υπομονή επί χρόνια έγιναν οι διαπραγματεύσει, οπότε πρόκειται τελικά για μια στεγανή συμφωνία σφαιρική με την οποία και συμφωνεί πρόκειται να έχουμε απτά κέρδη ε, εμείς και οι ευρωπαϊκέ εταιρείε δηλαδή. Και αυτό αφορά επίση και τους δασμούς. Οπότε μόλι τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία πρόκειται να έχουμε 500 εκατομμύρια ετησίω ω κέρδος ή ωφέλεια. Πρόκειται για την άρση των δασμών. Ε, επίσης θα ωφεληθούν και οι υπηρεσίες, θα ωφεληθούν οι επενδύσεις, θα αποκτήσουν πλεονεκτήματα οι ευρωπαϊκές εταιρείε. Όσον αφορά την έγκριση των επενδύσεων του στον Καναδά, ε, επίσης ο κ. Κοβατσέπ τονίζει ότι στη ΣΕΤΑ προβλέπεται και μια δυναμική διαδικασία για αναγνώριση κάποιων ε, δεξιοτήτων επαγγελματικών όσον αφορά το εξωτερικό σε διάφορου κλάδου. Ε, επίσης τονίζει ότι οι Ευρωπαίοι επαγγελματίε επίση και οι συνεργάτε των ε, φορέων μα των νομικών προσώπων μπορούν να δουλέψουν σε άλλη πλευρά του Ατλαντικού για άλλο οργιασμό των ευρωπαϊκών εταιριών και έτσι να τη βοηθήσουν τη δραστηριότητά τους αλλά και αντίστροφα για του ε, Και έτσι θα είναι δυνατόν να παρασχεθούν οι σχετικές υπηρεσίες και αυτό θα αφορά και επίσης κάποιες ε, κρατικές προμήθειες ε, σε κρατικό επίπεδο επομένω, αλλά και πιο κάτω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιου είδου δημόσιε συμβάσει σε σημαντικού ε, τομεί όπω φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό, εταιρείε υδάτων, σιδηρόδρομοι, αστικέ συγκοινωνίε. Και από ό,τι θα έχουμε καινούργιε ευκαιρίε, λέει ο κύριο Κόβατσεφ και για τον αγροδιατροφικό τομέα και ταυτόχρονα πρόκειται να προστατευθούν τα σημεία που μας ενδιαφέρουν, καινοτομία και θα κατοχυρώνονται και τα ατομικά δικαιώματα. Τα κοινωνικά πρότυπα, το περιβάλλον επίσης. Τέλος, είναι βούλος ο κ. Κόβατσεφ και ως τιούτος λέει ότι τελικά Επιτέλους κλείστηκε αυτή η συμφωνία γιατί έτσι πια δεν θα απαιτούνται βίζες στα διαβατήρια για Βούλγαρους και Ρουμάνους. Από 12 του 2017 μάλλον. Οπότε, επαναλαμβάνω ότι συμφωνεί 100% με το κείμενο του κύριου Τάνακο, κύριο Σκόβατσεφ. Οπότε και προτείνει το να ψηφίσουμε υπέρ της έγκρισης της συμφωνίας τα... για τους σοσιαλδημοκράτες, ο κύριος Λόπες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γρουπο, Μιλώ εξ ονόματος της ομάδας μου, αλλά να σας εξηγήσω τη θέση του Αντώνιο Παντζέρη, που είναι αρμόδιος για αυτό το θέμα. Μετά από όλη αυτή τη δουλειά που έχει κάνει. Και μιλώ εξ ονόματός του, λοιπόν, για να σας διαβιβάσω την άποψή του. Κολλείται δυστυχώς και αποσιάζει σήμερα. Πρώτον, ο κύριο Παντζέρη αυτό που επιθυμεί είναι να διαβιβάσει τι ευχαριστίες του στον κύριο Τάνοκ για τη δουλειά του, αλλά ομολογεί ταυτόχρονα ότι είναι δύσκολο ένα σκιώδη συζητητή για μια τέτοια γνωμοδότηση να μην μπορεί να κάνει τροπολογίες. Και μοναδική λύση είναι να το δεχτούμε ή όχι. Είναι λίγο ασπρομαύρο αυτό. Ο κύριος Παντζέρη θα επιθυμούσε να αλλάξουν αυτοί οι κανόνες και να μην έχουμε τέτοιου είδους νομοδοτήσεις ε, με ένα τέτοιο ναι ή όχι. Δεν πρόκειται να γνωμοδοτήσει ο κύριος Παντζέρη για τη ΣΕΤΑ εάν δεν ξέρει τι θα κάνει το Κοινοβούλιο. Ποια θα είναι η συμφωνία. Γίνονται και διάφορες ε, ερμηνευτικές δηλώσεις για τα διάφορα στάδια και τις νομοδοτήσεις που θα ακολουθήσουν. Υπάρχει κίνδυνος να μην ψηφιστεί μια συμφωνία ή να ψηφιστεί μια συμφωνία με πολλά ε, αφήσιμα ε, εδάφια. Μετά από όσα έγιναν στη Βουλή της Βαλονίας, υπήρξε μια στασιμότητα ε, που μπορεί να οδηγήσει το Βέλγιο να προσφύγει στο δικαστήριο για να ελέγξει κατά πόσο συνάδει η συμφωνία αυτή με το κοινοτικό και εκτιμένο ή την Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη. Ο κύριος Πανσέρη λοιπόν θα ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα έτσι ώστε κάπου να συμπεριληφθεί ε, και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο πλευρό του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Μπίχνερ από τους Πρασίνους, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως είμαστε όλοι υπέρ της ε, αύξησης ε, του δημερούς εμπορίου με τον Καναδά και θέλουμε ε, και να μειωθούν και οι δεσμολογικοί φραγμοί, αλλά θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Δηλαδή, η εξουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ε, προβαίνει στη σύναψη εμπορικών συμφωνιών και η ίδια η δυνατότητα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωση, να συνάπτει τέτοιου είδου συμφωνίας ε, ρυθμίζονται στο άρθρο 207 της συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Αυτό όμω αφορά τις εμπορικές συμφωνίες αμυγό. ενώ εδώ έχουμε να κάνουμε μια παρέμβαση μέσω τη ΕΤΑ ε, στην διοικητική αλλά και δημοκρατική δομή των κρατομελών. Σας υπενθυμίζω δηλαδή ότι η νομοθεσία παραμένει περιορισμένη Δηλαδή περιορίζεται από τι, από την προϋπόθεση ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν αχρίαστα εμπόδια σε ό,τι αφορά το ελεύθερο εμπόριο. Και ακριβώς αυτά τα περιτά εμπόδια, αυτά τα αχρίαστα εμπόδια είναι που δημιουργούν όλο το ε, πρόβλημα γιατί στο αγγλοσαξονικό δίκαιο ε, τη χάνει άλλη ερμηνεία από, από το πυρωτικό ευρωπαϊκό δίκαιο αυτό ο όρο. Αλλά ό,τι και αν αυτό ισχύει, ε, όπω και αν αυτό ερμηνευτεί, δεν μας ενδιαφέρει. Εκείνο που μα ενδιαφέρει είναι ποιε θα είναι οι αποφάσεις που θα λαμβάνουν τα διατηρητικά δικαστήρια. Και αυτό έχει να κάνει με τις ε, δυνατότητες ε, και τα δικαιώματα των κρατών μελών. Τα επενδυτικά δικαστήρια τα οποία προβλέπονται στο πλαίσιο αυτή τη συμφωνία δεν πληρούν ούτε τα ελάχιστα ε, ε, πρότυπα τα οποία θα πρέπει να πληρούν για παράδειγμα τα δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, που από και Οπότε είδαμε ότι οι εταιρείε Bagger και BASF χρηματοδότησαν ε, μαζικά την υποψηφιότητα του κυρίου Τραμπ, ο οποίος ακριβώς έχει ταχθεί κατά τη σύναψη τέτοιου είδους συμφωνιών. Αυτό μα δείχνει το τι ακριβώς συμβαίνει. Ε, νομίζω πως θα πρέπει σε γενικές γραμμές να πούμε ναι, επίτευξη του εμπορίου φυσικά και ε, ενίσχυση του εμπορίου, αλλά από εκεί και μετά είμαστε κατά ε, της εμπλοκής στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών μελών και γι' αυτό θα καταψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία ο κύριος ε, Μάριο Πετριτσόνε έχει ε, το λόγο από την πλευρά της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου και από την Ειδική ε, Μονάδα της Διεύθυνσης Εμπορίου. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. με χαρά μου βρίσκομαι σήμερα εδώ για να δώσω κάποιες διευκρινήσεις. δεν θα πω πολλά. Νομίζω πως ο εισηγητής περιέγραψε με ακρίβεια τη συμφωνία, οπότε δεν θα επισέλθω στο ζήτημα της οικονομικής αξίας αυτής της συμφωνίας. Απλά θα ήθελα να πω το εξή. Συχνά γίνεται μια ανάλυση της με βάση τη γενική οικονομική ε, σημασία αυτής της συμφωνίας σε ό,τι αφορά ε, την, ε, το σχετικό μέγεθος των δύο συμβαλωμένων μερών. Και νομίζω πως δεν είναι σωστή η οπτική γωνία. Δηλαδή, αν δούμε δηλαδή ποιος θα είναι ο αντίκτυπος σε σχετικό επίπεδο προφανώς 20 ε, φορές μεγαλύτερη είναι η ευρωπαϊκή οικονομία από αυτή του Καναδά. Αλλά ε, ας δούμε γενικότερα ότι πρόκειται για αύξηση του εμπορίου και από εκεί και μετά η εξάλληψη των ε, εμπορικών φραγμών, για παράδειγμα των ε, δασμών, μπορεί να δώσει την δυνατότητα και σε αυτή τη χώρα να, να δημιουργήσει περισσότερε θέσει εργασία ε, και να αυξήσει το εμπόριο. Μετά από εκεί και μετά, ε, όπω ισχύει από την. Ε, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας δεν μπορεί να εφαρμοστεί καμία συμφωνία προτού δώσει τη συμφωνία του γνώμη το Κοινοβούλιο, δηλαδή έχει συμφωνηθεί προσωρινή εφαρμογή αλλά χωρίς την συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ισχύει τίποτα. Από εκεί και μετά μια διευκρίνηση σε ό,τι αφορά τις διάφορες ερμηνείες ε, που έχουν ε, γίνει αυτές τι συμφωνίες και τις διάφορες διακηρύξεις που έχουν γίνει σε σχέση με αυτή τη συμφωνία και οι ερμηνείες πραγματικά είναι αναρρύθμιτες. Ε, νομίζω τα όσα έγιναν στο επίπεδο δηλαδή του ζητήματος που προέκυψε με τη Βαλονία και στο των συζητήσεων που έγιναν με άλλα κράτη-μέλη, ε, θα πρέπει να πούμε ότι δεν άλλαξε το περιεχόμενο της συμφωνίας. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες ρήτρες οι οποίες θα ενεργοποιούνται αν θέλετε νωρίτερα και ε, θα δώσουμε και συγκεκριμένες ε, διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά αυτή την αναθεώρηση και το προς τα που θα, προς θα κατευθυνθεί. Ε, δηλαδή σίγουρα και ο Καναδάς θα συμφωνήσει με αυτές τις με αυτές τις συμπληρωματικές με βάση δηλαδή και τις συζητήσεις που κάνουμε κατά του τελευταίους μήνες. Οπότε η Επιτροπή από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επί του συγκεκριμένου συστήματος, ε, ακολουθώντας την κατεύθυνση που ήδη αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής. Δηλαδή μια κατεύθυνση η οποία ήδη προβλέπεται από το πνεύμα της συμφωνίας και η οποία ήδη έχει συμφωνηθεί με την κυβέρνηση του Καναδά. Η, το, η κυβέρνηση της Βαλωνίας από εκεί και μετά μπορεί να ζητήσει από την κυβέρνηση του Βελγίου να ζητήσει μια γνωμοδότηση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τη συμβατότητα αυτών, του αποτελέσματος δηλαδή αυτής της συμφωνίας ε, με τι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εμεί είμαστε πεπισμένοι ότι δεν θα, δεν θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί δεν θα προχωρούσαμε στη σύναψη μια συμφωνία αν είχαμε οποιαδήποτε αμφιβολία σε ό,τι αφορά τη συμβατότητα με τι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν έχουμε και καμία αντίρρηση στο ένα κράτο μέλο να απευθυνθεί στο δικαστήριο για να ζητήσει διευκρίνηση σε ό,τι αφορά αυτή τη συμβατότητα. Άρα δεν πρόκειται εδώ για να ε, ζήτημα ε, αμφισβήτηση τη συμφωνία. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση ό,τι αφορά τη συμβατότητα. Δηλαδή, εάν πει το δικαστήριο ότι υπάρχει ζήτημα συμβατότητα με τη συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να ε, αναλάβουν τι σχετικέ δράσει. Αυτά από την πλευρά μου. Ευχαριστώ πρώτα. Ευχαριστώ. Κύριο Σκέλα, τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. General observations να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον συνάδελφο Τάνοκ για το εξαιρετικό του κείμενο. Uh, ε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι εκφράζονται έτσι γνήσια τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συμφωνία ΣΕΤΑ θα συνεισφέρει τα μάλα στη δημιουργία αλλά και ενίσχυση ε, παγκοσμίων προδιαγραφών για το εμπόριο για τον 21ο αιώνα με διαφάνεια και σαφήνεια, διότι ο Καναδάς υπήρξε στρατηγικός μας σύμμαχος εδώ και μία 20 ετία. Είναι και σύμμαχός μας γενικότερα στη διεθνή πολιτική. Και ελπίζω η συμφωνία ΣΕΤΑ να βοηθήσει να εστιαστεί η προσοχή και πάλι στις διατλαντικές σχέσεις και να ξεφύγει από τον ειρηνικό που έχει ε, μετατοπιστεί. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε και ένα μόνιμο δικαστήριο επενδύσεων που θα είναι ένας μηχανισμός προσφυγών. Και δεν θα πρέπει να υποτιμούμε ή να παραμελούμε το γεγονός ότι με τη Συμφωνία ΣΕΤΑ τώρα έχουμε μια νέα σχέση στρατηγικής εταιρικής έτσι, συμφωνίας με τον Καναδά. Και χαίρομαι που τρεις, μάλλον τέσσερις μεγάλες πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο υποστηρίζουν την προσπάθεια αυτή και τη συμφωνία. Και εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνάδελφο Τάνοκ και σε όλους μας. Ευχαριστώ. Any other, uh, Άλλος συνάδελφος? Θέλει να λάβει το λόγο, όχι από ό,τι βλέπω. Ο εισηγητής και πάλι για να ολοκληρώσει, για να κλείσει. Θέλω μόνο να σχολιάσω κάτι. Μήπως ε, δεν κατάλαβα κάτι από τη διερμηνία. Όταν μίλησε ο σοσιαλιστικής συνάδελφος εξ ονόματος του κυρίου Παντζέρη, είπε ότι λυπάται από το γεγονός ότι δεν μπορεί να, να τροποποιήσει τη γνωμοδότησή μου. Όχι τη γνωμοδότησή μου, τη συμφωνία. Η δική μου γνωμοδότηση δέχεται τροπολογίες. Ούτε η δική μου. Ναι, είναι. Η γνωμοδότηση βέβαια επιδέχεται τροπολογίε. Το δικό μου κείμενο, ναι. Προφανώ δεν μπορεί κανεί να τροποποιήσει τη συμφωνία, τη συνθήκη που είναι η σύμφωνη γνώμη, ναι ή όχι. Αν υπάρχει τίποτα στη δική μου γνωμοδότηση που να μην του αρέσει, θέλει να προσθέσει κάτι με χαρά ε, να τι υποβάλει και εγώ θα τι διαβάσω με μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Πριν κλείσουμε αυτό το θέμα, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι υπάρχει προθεσμία για τροπολογίες αύριο 15 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Και όπως είπε και ο συντάκτης νομοδότησης, μόνο ε, τροπολογίες που μπορεί κανείς να υποβάλει είναι απόρριψη, ε, να μην δοθεί σύμφωνη γνώμη. Ε, το επόμενο θέμα έχει προβλεφθεί για τις 5.30 και χρειάζεται απαρτία για να ψηφίσουμε, γιατί προς το παρόν μόνο ποδοσφαιρική ομάδα φτιάχνουμε. Μικρή διακοπή πέντε λεπτών. Ladies and gentlemen, take your seat. We are... Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι για να συνεχίσουμε. Ladies Κυρίες και κύριοι, συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Ε, περνάμε λοιπόν στο σημείο 6 της ημερήσιας ε, διάταξης, ε, δηλαδή εκλογή του τετάρτου αντιπροέδρου. Όπως γνωρίζετε, ο προηγούμενος αντιπρόεδρος, κ. Μάκοβιτς, κατέστησε αντιπρόεδρος στη δική του χώρα, οπότε θα πρέπει να εκλεγεί τώρα ο αντικαταστάτης του. Έχουμε νομίζω τώρα πλέον Ολομέλεια εδώ τον απαραίτητο αριθμό ε, το μελών, δηλαδή 18 μέλη. Έχουμε περισσότερα από 18 μέλη αυτή τη στιγμή μεταξύ μόνο οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκλογή. Θα ήθελα να σας ζητήσω όσοι θέλετε να θέσετε την υποψηφιότητα, Κύριος Γκάλ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, από την πλευρά του ΕΛΚ. Θα ήθελα να προτείνω την κυρία του Μπρεβοσβίτσα για την θέση της τετάρτης αντιπρόεδρου σε περίπτωση που εκλεγεί θα ήθελε να αποδεχθεί αυτή την εκλογή της. Απλά αυτή τη στιγμή είναι ακόμα στο αεροδρόμιο του Μονάκου και δεν μπορεί να συνεχίσει. Ναι, ε, ε, πληρεί όλα τα κριτήρια η εν λόγω υποψήφια. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Εάν όχι, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιος είναι υπέρ της εκλογής της κυρίας Σουίτσα. Thank you very much. Καλώς, νομίζω πως η απάντηση ήταν ε, σαφής, οπότε συγχαίρουμε εν τη απουσία της ε, την κυρία Σούτσα. Οπότε θα τη συγχαρούμε και προσωπικά την επόμενη φορά που θα είναι εδώ μαζί μας. Οπότε κλείνουμε και με αυτό το σημείο και περνάμε στην ψηφοφορία σε σχέση με την ε, έκθεση σε ό,τι αφορά την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είναι μια αρκετά μακροσκελή ε, διαδικασία ψηφοφορία και ο σχετικό κατάλογο. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω τη συνεργασία σα. Δεν ξέρω αν ο εισηγητή, ο κ. Βαντικό θα να πάρει το λόγο για να πει τίποτα. Ε, θα ήθελα απλώ να ευχαριστήσω όσου ε, όλου συνέβαλαν στην κατάρτιση αυτή τη έκθεση. Δεν θα μακρηγορήσω γιατί έχουμε πράγματι μια, ένα μακροσχέλη κατάλογο ψηφοφορία. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ. Εκτιμούμε λοιπόν την παρέμβασή σα. Σα παρακαλώ να ετοιμάσετε τι ε, κάρτε ψηφοφορία σα εδώ. Και α ξεκινήσουμε με τη συμβαστική τροπολογία 19 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 20. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. Τροπολογία 191. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτω. Συμβαστική τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 197. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 22. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 23. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 207. Ψήφιπερ Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε τη 207. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τροπολογία 207. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Vote is closed. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 208 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε. Ελέγχουμε τη 208. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επόμενη είναι συμβαστική τροπολογία 24. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 221 ψήφι κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 222 ψήφι υπέρ. μηματική λοιπόν ψηφίζουμε επί του πρώτου ε, μέρους της 222 ψήφι κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μέρος δεύτερο ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται. 223 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 224 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 26 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 231. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ...237 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 27 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 28. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 29. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 248 ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 30. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 31. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 266. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 270 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική, 271 δεν είναι συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 32 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 275 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 276 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 277 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 278 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 33 Συμβαστική τοπολογία 33, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 284, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 285 ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 286 ψήφι υπέρ κατά αποχές θα, θα ήθελα να ελέγξουμε τη 286 άρχεται η ψηφοφορία Vote is closed. Πέρασε ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 293. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 294. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 295. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. τροπολογία 296. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 297 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 298 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 299 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 300 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 301 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 302 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 303 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 304 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 305 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 307 τσεκ φωνές από κάτω. Την 306 λοιπόν θέλετε να ελέγξουμε. Παρακαλώ, ηλεκτρονική επαλήθευση. Συντροπολογία 306. Αρχίζει και τελειώνει η ψηφοφορία. Απερίφθη. Με μικρή διαφορά. Η τροπολογία 307. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 308. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 309 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 310 υπέρ κατά αποχές Εδώ θα ήθελα ένα έλεγχο παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία γιατί δεν είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Πέρασε. Απορρίπτεται, όντως. 311 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 312 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τσεκ, καλώς. Ελέγχουμε την τροπολογία 312. Vote is open. Vote is Αρχίζει και δηλώνει η ψηφοφορία. Sorry, αλλά είχε απορριφθεί σαφώς. Την άλλη φορά παρακαλώ πριν ζητήσετε τσεκ ε, να το ξανασκεφτείτε. Ε, η συμβαστική 37. Τι έγινε, 3 13 καμία τροπολογία. 3-13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, τώρα θέλει έλεγχο όμως. 313. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρασε. Η συμβαστική 37 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Η συμβαστική 38 υπέρ. Κατά αποχές Νομίζω ότι είχε απορριφθεί, αλλά ας την ελέξουμε παρακαλώ, τη συμβαστική τροπολογία υπερθμών 38. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Α, είχε εγκριθεί. Η τροπολογία 326. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 327 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 328 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 329 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική. 39. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 347 ψηφί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 40 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 349. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 350. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 351. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 353. Υπέρ, κατά, παπουχές εγκρίνεται. Η 355 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 356 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 358 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 360 υπέρ. 61 συγγνώμη. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα η 360 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Η 359 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Η 362 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα έχουμε χωριστή ψηφοφορία στην 363. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και δεύτερο τμήμα πάντα στην 363 υπέρ κατά αποχές απορρίψεται. Τώρα θα ψηφίσουμε τις επόμενες τροπολογίες 364, 65 και 66 που είναι ταυτόσιμες. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 367 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 368 υπέρ. Κατά. Αποχές Έλεγχος παρακαλώ, ότι 368 τώρα ελέγχουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 369 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 370 υπέρ κατά αποχές εδώ χρειάζεται έλεγχο. Ηλεκτρονική επαλήθευση της ε, τροπολογίας 370. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 41. Ψήφι Π. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Με 385 ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Συγγνώμη, συμβαστική τώρα 42 ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 43 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 406 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική όχι, τροπολογία 407 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 408. Ο πρόεδρος λέει συμβαστική, κανονικές τροπολογίες. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 409 κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Νόου, no, φωνές από κάτω. Ας το ελέγξουμε λοιπόν. Συμβαστική 44. Πέρασε. Μάλιστα, είχε εγκριθεί. Συμβαστική 45. Υπέρ, κατά, αποχές, Τώρα χρειάζεται έλεγχος εδώ. Ευχαριστώ. Πέρας. 44-9 εγκρίνεται. Uh, amendment 422. Ε, Κατά. Αποχές. I can make Και απορρίπτωται. Μπορεί να κάνω γράφη, αλλά ούτε εσείς με βοηθάτε, λέει ο κύριος Κούκαν. Κάνουμε ηλεκτρονικό όσον αφορά το 422. Ψηφίζομαι. Πέρας. Α, εγκρίθηκε. 423. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 424 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 425 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 426 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 427 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 429 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 430 υπέρ κατά α, αποχές εγκρίνεται 431 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για το 431 ψηφίζουμε πέρα ψηφοφορίας απορρίπτωται 432, 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 433. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Αφορά την 433. Πέρασε ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 434 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 440 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 441 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 449 χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα 449 υπέρ κατά αποχές τηλέφωνο φωνάζει κάποιο γιατί κουδουνίζει τηλέφωνο. Κάνουμε το ηλεκτρονικό του με το 349, λέει ο κύριο Κούκαν. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφορία. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα της 449. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Δεν χρειάζεται ηλεκτρονικό έλεγχος. Πλάκα κάνετε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην συμβαστική 49. Υπέρ, κατά. Α, αποχές. Ε, εγκρίνεται. Συμβαστική 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, εγκρίνεται. 51 in favor. Συμβαστική 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Abstentions carried. Αποχές και εγκρίνεται υπέρ 52. Τροπολογία 463 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 464 υπέρ. όχι, όχι, συγγνώμη. Συμβαστική 53, διορθώνει ο πρόεδρος, 53 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται η συμβαστική 53. 469 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 470 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 471 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Νομίζω ότι απορρίφθηκε πάντως. Ψήφιζουν. Πέρα της εφορίας. Όντως απορρίπτεται 472 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 473 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτωτα. Συμβαστική 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 477. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτωτα. Ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. 477. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Όντως έχει απορριφθεί. 478. Κάτι λέει ο κύριος Στάνοκ εκτός μικροφώνου. Εγώ θα ψήφιζα υπέρ, λέει ο κύριος Στάνοκ, κάτι τέτοιο. Charles, sorry, it would have been... Συμπάθαμε, Charles, αλλά το σωστό είναι να μου το έλεγε στην αρχή, στην αρχή της ψηφοφορίας. Αυτό δεν είναι συμπεριφορά κυρίου λέει ο κύριος Κούκαν. Α, τώρα κατάλαβα, λέει ο κύριος και να λαμβανόταν υπόψη η ψήφος μου, δεν θα άλλα το αποτέλεσμα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Εντάξει, Τσάλ, θα καταμετρηθεί η ψήφος, θα καταχωρηθεί τέλο πάντων. Άρα εγκρίνεται. Ήταν κρίσιμη ψήφος. Πάμε τώρα στο 478, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για το 478. Πέρασε ο φορείος. Εσύ, Τσάλς, τι ψηφίζεις αυτή τη φορά. Εκτός μικροφώνου, τα σχόλια. Άρα απορρίπτεται. Σύμβαση 55. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 493 υπέρ κατά αποχές νομίζω εγκρίνεται αλλά ας κάνουμε έλεγχο 493 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά πέρας εγκρίνεται 498 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 499 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 500 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 501 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος για την 501 Ψηφίζουμε πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Όπως σας είπα. 502. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Από όσους ψηφίσαν τέλο πάντων. 505 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. 507. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 508 υπέρ κατά α, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 512 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 513 υπέρ κατά αποχές. Λειτουργικός έλεγχος για το 513. Ψηφίζουμε πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 60. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 500. 91 Συγγνώμη, 519. Υπέρ κατά αποχές το 519. Όμως σας γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος δια το 519. 519 μάλιστα. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Charles, you voted against, yes? Charles ψήφισε κατά, έτσι, καλώς. Άρα λοιπόν απορρίπτεται σε αυτήν την περίπτωση. 520. Η απόφαση μου ήταν ότι θα ληφθεί υπόψη η ψήφος συνάδελφου. 520 λοιπόν ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την τροπολογία 520, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρασε τη ψηφοφορία και απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 521, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 522 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 61, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Όχι. Σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας, γιατί έτσι όπως είδα εγώ ήταν απορρίφθηκε, αλλά εντάξει. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τη συμβαστική τροπολογία 61. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η επόμενη είναι η συμβαστική τροπολογία 62. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική ή μάλλον κανονική 547 ψήφι υπέρ. 548 συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 548 το Τροπολογία 548 λοιπόν, η ψηφοφορία. Λοιπόν, λίγε ψήφοι ακόμα. Πέραση τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται λοιπόν. 549 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 550 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 551 υπέρ, κατά απουσίας απορρίπτεται συμβαστική 64 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται συμβαστική 65 υπέρ κατά απουσίας εγκρίνεται συμβαστική 66 υπέρ κατά απουσίας εγκρίνεται τροπολογία 567 μαζί με την 568 για την ε, ταυτόσημα ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 68 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 593 598 ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται Ελέγχουμε για αυτές τις τροπολογίες 593 598 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. 599 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 600 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 600. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της φοβορία. Εγκρίνεται. 601 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 602 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 603 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 604 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 605 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 606 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 607 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε. Την 607 πάντα. Ψήφι υπέρ. Ε, συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. εγκρίθηκε. 608 τώρα. Ψήφι πέτ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε και αυτήν. Ελέγχουμε την τροπολογία 608. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 609 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 610 υπέρ, κατά, αποχές να ελέγξουμε. την 610. Πέρας λοιπόν της ψηφοφορίας και εκρίθηκε. 612 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 613 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 614 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 615 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 616 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 617 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 620 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 623 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 624 υπέρ κατά αποχές Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 624 πέρας φυσφοφορίας και εγκρίνεται. Συμβαστική τοπολογία 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 628 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 631 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 71 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 637 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 638 υπέρ, κατά αποχές. Να ελέγξουμε την 638. πέραση τη ψηφοφορία εγκρίνεται. 639 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 72 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εξα... Συμβαστική 73 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε τη συμβαστική τροπολογία 73. Πέρας της Εγκρίνεται. 656 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 665 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε την 665. Πέραση της φοβορίας Απορρίπτεται. 666 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Όχι, δεν συμφωνείτε, να ελέγξουμε την 666. Πέρας της φοφορίας απορρίπτεται. 667 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 668 σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε επί του πρώτου τμήματος, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εάν δεν διαμαρτυρηθείτε πολύ, ο πρόεδρος και περνάμε οπότε δεν ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα συμβαστική 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 675 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 676 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 677 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 687 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 600 687 λοιπόν αλέξουμε την 687 ηλεκτρονικά πέρασε η ψηφοφορίας Εγκρίνεται λοιπόν Περνάμε στην 688 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 76 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ...708 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, ...709 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 710 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα έλεγα 711 υπέρ κατά αποχές απορρίπτε 714 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όχι δεν συμφωνείτε 714 λοιπόν ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 714. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 715 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 716 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 717 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 718 υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 719 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 720 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 721 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 77 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 730 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 731 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 732 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 733 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 734 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε την 734. ψηφοφορίες. Απερίφθη. Προχωρούμε. Τροπολογία 735 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 736 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 737 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 78. Τσεκ. Ωραία. Ε, ελέγχουμε λοιπόν την 737 ηλεκτρονικά. Και όντως είχε απορριφθεί. Δίκαιο είχατε. 78 λοιπόν συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 740 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 741 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 742, όχι, 741. Την ελέγχουμε λοιπόν. Αρχίζει. The vote It was rejected. Απερίφθη. 742 in favor. 742 υπέρ, κατά. Αποχές με την ίδια πλειοψηφία. Απερίφθη. 7.43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7.44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7.45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7.46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7.47 υπέρ κατά αποχές. Αυτό θέλει έλεγχο παρακαλώ. 7.47 The is closed. Πέρασε. Ο Τσάρλς Τάνοκ έχει την αποφασιστική ώρα ψήφο. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. 748. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ε, κοιτάξτε πόσο σημαντικός μπορεί να είστε ε, αν ξεχνάτε την κάρτα ψηφοφορίας. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, 7.50 ναι, έχουμε κατά τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7.51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7.52 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 7.53 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 7.54 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική 79 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Η 7.61 υπέρ. Κατά. Απόχες Ας την ελέγξουμε λοιπόν. 761 ηλεκτρονικός έλεγχος. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Απέριφθη. 763 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 762 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 765 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 767 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 771 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 777 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 778 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 779 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 780 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 781 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 782 τσεκ την 781 ηλεκτρονικά λοιπόν Πέρας. Περιμένω να μου στήσετε συγγνώμη. Όχι, όχι. Εγώ ζητώ συγγνώμη όταν κάνω λάθη, θα έπρεπε να κάνετε και εσείς το ίδιο. 782 είπε. Είπα sorry, λέει η κυρία Βερζιά. Είπα sorry. Α, συγγνώμη που δεν είπα ότι λυπάστε. Ωραία. 782 είπε. Κατά αποχές έλεγχος τώρα την 782. Πέρασε. Sorry, τώρα εγώ λέω πέρασε. Τρεις φορές. 783 είπε. κατά, αποχές απορρίπτεται. 784 Τώρα θέλετε έλεγχο στην 783. Πάμε λοιπόν. Ηλεκτρονική απολύθευση. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 784 επέ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 785 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 786 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 788 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 789 υπέρ κατά αποχές Ας την τσεκάρουμε αυτή 789 ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Πέρασε. Απερίφθη. 790 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 791 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 792 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στην 793 τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. No. Ελέγχουμε λοιπόν το δεύτερο τμήμα της 793 ηλεκτρονικά. Απερίφθη λοιπόν. Η τροπολογία 794 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 802 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 803 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 804 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 805 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 806, 807, 808 μαζί όλες αυτές υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται η συμβαστική 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Οι 8-18, 19, 8, 28, 22, 21 και 23. Όχι, η 821 έχει αποσυρθεί. Όλες τις άλλες μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτονται. Τροπολογία 824, 23, συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα έχουμε τις τροπολογίε 824, 825. Όχι, πάμε στην 839. Καλύπτονται από προηγούμενο συμβιβασμό. 840, 41, 43 και 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Όχι. Yes. Εγώ από εδώ το είδα για απόρριψη πάντως. 8, 45, 46, 47 υπέρ κατά αποχές τώρα θέλει έλεγχο. Παρακαλώ αρχίζει ηλεκτρονική απολύθευση. Πέρασε. Απερίφθη. Συμβαστική 83 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 84 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 854 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η, η τροπολογία 855 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. συμβαστική 85 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 861 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 863 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 864 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 865 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 866 υπέρ κατά αποχές εδώ θέλει έλεγχο 866 αρχίζει ο έλεγχος πέρας εγκρίθηκε λοιπόν τώρα έχουμε την τροπολογία 47 Ψηφίπε. κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60 υπέρ κατά Α, έλεγχος. 60. Ε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Μικρή διαφορά. Κύριε Τάνοκ, που θα γυρεί πλάστιγκα. Κατά Όχι, εγκρίθηκε. Όχι, καθόλου, ισοψηφία. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι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 κατά αποχές εγκρίνεται. Η ε, τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 90 υπέρ κατά αποχές. Ας την ψηφίσουμε την τροπολογία 90 παρακαλώ. Πέρας. Απερίφθη. Συνεχίζουμε. Η τροπολογία 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, τα τμήματα 104 το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 112 και 113 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μαζί 112-113 ηλεκτρονικός έλεγχος και των δύο αυτών τροπολογιών. Πέρας. Εγκρίθηκαν. Η τροπολογία 114 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέ κατά αποχές απορρίπτεται. 119 υπέ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τροπολογία 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται χωριστεί στην 147 τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Συμβαστική 16 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. και 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 158 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 161 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 162 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική 18 υπέρ, κατά αποχές. α, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ, συμβαστική 18. The Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 169 υπέρ. Κατά. αποχέ. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν την 169.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 ε, αποχές 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται συγγνώμη 16 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 16 Ελέγχουμε λοιπόν τροπολογία 16 ηλεκτρονικά. The vote is closed. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 22 λοιπόν ηλεκτρονικά. Πέραση της φουφορίας εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική λέει ο 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την τροπολογία 35. The vote is closed. Εγκρίνεται λοιπόν. Περνάμε στην 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Περνάμε στους ψήφους Ντέβε. No, no, objection, no objections to the Δεν υπάρχουν εδώ αντιρρήσεις. από το ΔΕΒΕ 3 λοιπόν έως το ΔΕΒΕ 15 συνολικά ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ και περνάμε πάλι στην ομαδική για τις Όχι, δεν συμφωνούμε όλοι. Οπότε θα πρέπει να τις ε, ψηφίσουμε μία προς μία. ΔΕΒΕ 1 υπέρ, κατά, DV10, DV10 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. DV, όχι. 5, 5, 10. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. για την Πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 513 εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 λοιπόν. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την ΦΕΜ 27. Πέραση εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Να σε ελέγξουμε την ΦΕΜ 75 ηλεκτρονικά. Πέρας της πληροφορίας πράγματι απορρίπτεται. Για τις επόμενες τώρα θα ήθελα να προτείνω unblock από την 1 έως την 91. Τροπολογίες λοιπόν φέμ 1 έως 91 κατά αποχές. Σας ευχαριστώ. Όλες αυτές λοιπόν οι απορρίφθηκαν. Και τώρα περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σχέδιο ε, του ψηφίσματο όπω αυτό τροποποιήθηκε με τι τροπολογίε. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Το ψήφισμα λοιπόν εγκρίνεται. Τα συγχαρητήριά μα στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνουν μια ψηφοφορία. Η επόμενη συνάντησή μας είναι στις 24 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο και μετά στις 29 Νοεμβρίου. Σα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Πέρα συνεδρία